works this way. Okay, right. If uh, everybody is ready, we'll, we'll start because. Uh... Αν είστε έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε. Γιατί θέλω να είμαστε εντό χρονοδιαγράμματο. Πρώτα απ' όλα έχουμε την υιοθέτηση της μέσης διάταξης Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ωραία. Θα Κάνουμε όλες τις ανακοινώσεις αύριο. Και έτσι το μοναδικό θέμα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι ο νομισματικός διάλογος με τον κύριο Μαριο Ντράγκη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και μετά θα περάσουμε σε δεύτερη συνεδρίαση στη δημόσια ακρόαση με τον Μάριο Ντράγκη ως ε, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές ε, συνεδριάσεις προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα σταθμό, έναν βαθμό διάκριση μεταξύ των δύο. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον Μάριο για τις ενακτήριες παρατηρήσεις του και μετά θα περάσουμε στον γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων, ως ήχθιστε. Και τώρα έχουμε τον νέο μορφότυπο των ε, χρονοθερίδων 5 λεπτών. Αν δοθεί λοιπόν η ευκαιρία θα επανέλθετε. Αν δεν έχει, υπάρχει χρόνος, τότε δεν θα συμβεί αυτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νοσμικών Υποθέσεων, είναι με μεγάλη μου ευχαρίστηση που επανέρχομαι εδώ στο Κοινοβούλιο ενώπιον της Επιτροπής σας για την τακτική μας ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε πλέον μπει στο 2013 με ένα πιο σταθερό δημοσιονομικό περιβάλλον από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό επετεύχθη μέσω συγκεντρωμένων ε, προσπαθειών και αναδιαρθρώσεων των ε, κυβερνήσεων και των ε, κοινοβουλίων και αποφασιστικής δράσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Όμως πρέπει να καταληφθούν περαιτέρω από προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα ξεφύγει από αυτή την κρίση, θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη μεταξύ επενδυτών και πολιτών και θα επανεγκαθιδρύσει τη σταθερότητα και ανάπτυξη. Το Κοινοβούλιο έχει θεμελιώδη ρόλο να διδραματίσει σε αυτή τη ε, διαδικασία μεταρρύθμισης. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στην υιοθέτηση της ε, νομοθεσίας για ε, τον ενιαίο μηχανισμό επίβλεψης που είναι κρίσιμη σημασία για την διαδικασία αυτή. Σήμερα θα αναφερθώ πρώτα στις οικονομικές και ε, νομισματικές εξελίξεις ε, στην Ευρωζώνη από τον ε, Δεκέμβριο και μετά. Μετά θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα πιο συγκεκριμένα, τον αντίκτυπο του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων και την εγκαθίδρυση του ενιαίου επιπτικού μηχανισμού. Από τη τελευταία μας συνάντηση, το Κυβερνητικό Συμβούλιο έχει αφήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας στο 0,75% και για τις, ε, περιφερει... τις ε, οριακές ε, δραστηριότητες στο 1,5%. Η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα για το 2012. Η διαθέσιμη δείκτες δείχνουν περαιτέρω αδυναμίες στις αρχές του 2013, ε, καθώς έχει πέσει σε σημαντικό βαθμό η εσωτερική ζήτηση. Αυτό οφείλεται ε, στην αδύναμη ε, δραστηριοποίηση καταναλωτών και επενδυτών καθώς υποχωρεί και η εξωτερική ζήτηση. Η οικονομική αυτή αδυναμία στις αρχές του 2013 αναμένεται ότι θα ακολουθηθεί από ε, μια πολύ σταδιακή ανάκαμψη στη συνέχεια φέτος. Η ενίσχυση της ε, συνολικής και σφαιρικής ε, ζήτησης, η συνολική μας στάση σε ό,τι αφορά τα νομισματικά ζητήματα και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ε, στις χώρες Ευρωζώνης ε, θα μας βοηθήσουν ε, να λάβουμε και σημαντικές αποφάσεις και να στηρίξουμε την ανάκαμψη. Αν και ακόμα δεν υπάρχει πραγματική βελτίωση στην πραγματική οικονομία, ορισμένοι δείκτες μελετών μας έχουν επιβεβαιώσει προηγούμενες ενδείξεις σταθεροποίησης της και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης επιχειρήσεων και καταναλωτών, παρότι παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η βελτίωση όμω στη δημοσιονομική αγορά και στην εμπιστοσύνη από πέρσι το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντική. Σε ό,τι αφορά τα επιτόκητα, τα, τους, ε, τις αξίες πρέπει να ε, ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι στόχο πολιτική, αλλά είναι σημαντικό δείκτη για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών. Άλλη ένδειξη τη αυξημένη εμπιστοσύνη είναι η αποπληρωμή από του εταίρου μα. Ε, τις ε, πρώτες από τις ε, δύο τριετής ε, μακροπρόθεσμες επιχειρήσεις αναχρηματοδότησης που συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011 και τον Μάρτιο του 2012. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει τόσο ευεβαιότητα στις τράπεζες ό,τι αφορά τις χρηματοδοτικές προοπτικές σε σχέση με πέρσι. Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε εκ του σε την κατάσταση στην αγορά. Οι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προοπτικές για την Ευρωζώνη ε, παραμένουν και αφορούν ε, την χαμηλότερη από την αναμενόμενη ε, εσωτερική ζήτηση και τις εξαγωγές, την χαμηλή εφαρμογή των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρωζώνη, καθώς και γεωπολιτικά ζητήματα και ανισορροπίες σε, στις κύριες βιομηχανοποιημένες ε, χώρες μπορούν να έχουν αντίκτυπο στις εξελίξεις ε, στις χρηματαγορές ε, και στις αγορές εμπορευμάτων. Αυτό, αυτοί οι παράγοντες μπορούν να καθυστερήσουν την ανάκαμψη λόγω της καθυστερημένης αποκατάστασης εμπιστοσύνης. Η ετήσια, ο πληθωρισμός από το 2,5% τον Οκτώβριο πέρασε στο 2,2% τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και το 2,0% τον Ιανουάριο, ως είχαμε προβλέψει. Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί ε, σε κάτω από το 2% βραχυπρόθεσμα. Οι κίνδυνες ό,τι αφορά την, τις εξελίξεις των τιμών ε, θεωρούνται ως ε, εξισορροπημένοι πρόθεσμα με κάποιους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με τις ε, τιμές και τους έμεσους ε, φόρους καθώς και τις υψηλότερες ε, τιμές του πετρελαίου και έχουμε και άλλου είδους κινδύνους που απορρέουν από την, την πιο αδύναμη οικονομική δραστηριότητα και πρόσφατα την ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ. Η προσδοκίες σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη ε, παραμένουν ε, ε, συγγενείς ως προς το στόχο του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την επίτευξη του 2%. Σε ό,τι αφορά την νομισματική μας ανάλυση, συνδέεται με τη σταθερότητα των τιμών, το τίσιο ότι ίσως ο βαθμός αύξησης των ε, δανείων στον ε, ιδιωτικό τομέα παραμένει αρνητικός. Ε, σε μεγάλο βαθμό αυτή η αρνητική δυναμική αντικατοπτρίζει τον επιχειρηματικό κύκλο. Συνολικά, οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να είναι περιορισμένες στην επόμενη περίοδο. Και συλλέγοντα όλα αυτά τα στοιχεία, αυτό θα μα επιτρέψει να καθορίσουμε αντιστοίχω την νομισματική μα πολιτική. Α στραφώ τώρα στο άλλο ζήτημα που ε, θα μα απασχολήσει σήμερα, σε ό,τι αφορά τι επιπτώσει ε, του περιβάλλοντο χαμηλών επιτοκίων. Ο αντίκτυπο ε, τη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση στην οικονομία και στι εξελίξει των τιμών ήταν άνευ προηγουμένου αναγκαστήκαμε να λάβουμε μέτρα άνευ προηγουμένου ε, για να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε κινδύνους στη σταθερότητα των τιμών ε, σύμφωνα και με την εντολή μας. Πρώτον, μειώσαμε το βασικό ε, επιτόκιο στο 0,5% ποσοστό που προηγουμένως δεν είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν σε καμία από τις χώρες της Ευρωζώνης. Το επιτόκιο σε συγκεκριμένου τομεί όπω η αγορά Interbank είναι ακόμα χαμηλότερη, κοντά στο 0. δώσαμε στις τράπεζες απεριόριστη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε όλες τις χρηματοδοτικές δράσεις. Επεκτείναμε σημαντικά τον μέσο όρο ορίμανσης για αυτές τις δράσεις. Διευρύναμε τη βάση των εγγύσεων collateral. Και αυτή η διασφάλιση χρηματοδότησης των τραπεζών μπόρεσε να, να οδηγήσει στο να αποφύγουμε ασυμμετρίες και προβλήματα όσον αφορά αυτό το τομέα με πολύ σημαντικές επιπτώσεις εν δυνάμει για τη σταθερότητα των τιμών και για την απασχόληση και την ανάπτυξη επίσης εξίσου. Όλες αυτές οι αποφάσεις διασφάλισαν την σταθερότητα των τιμών και σταθεροποίησαν τις προσδοκίες ε, για τον πληθωρισμό κατά τη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής έκτακτης περίοδου. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει συνειδητοποιήσει τις προκλήσεις ε, που απορρέουν από μια παρατεταμένη περίοδο ε, χαμηλών επιτοκίων και ευρεία ρευστότητας. Α αναφερθώ σε τρεις κύριε προκλήσει. Η πρώτη, ότι αυτό θα μπορεί να έχει επιπτώσει στην δυνατότητα των εκταμιευτών και των επενδυτών για να σημειωθούν κέρδη. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, ονομαστικές ε, αξίες, όσον αφορά για παράδειγμα ασφαλιστικές εταιρείες ε, και συνταξιοδοτικά ταμεία. Ωστόσο διασφαλίζοντας την σταθερότητα των τιμών κατά την κρίση, η σταθερότητα αυτή των τιμών συνεισέφερε για ένα πιο σταθερό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Αυτό είναι κέριο ενδιαφέροντος και συμφέροντος ε, για τους ε, εκταμιευτές ε, και τους επενδυτές. Μόνο τότε μπορεί να υπάρξει, να υπάρξουν, να υπάρξει κερδοφορία όταν υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον. Δεύτερη πρόκληση. Η παρατεταμένη περίοδος χαμηλών επιτοκίων και ευρείας ρευστότητας διευκολύνει την μετακύληση των κινδύνων και έτσι πολλές φορές μπορεί να διατίθενται κονδύλια σε μη κερδοφόρες ε, δράσεις. Ε, με την πάροδο του χρόνου τέτοιου είδους εσφαλμένη τοθέτηση χρημάτων ε, θα υπονόμευε την παραγωγικότητα και θα μείωνε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τρίτη πρόκληση. Η παρατεταμένη αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει στο να υπάρξουν φούσκες στην αγορά στέγασης και σε άλλους τομείς. Όπως η κρίση κατέδειξε, η έκρηξη τέτοιων φούσκων έχει πολύ σημαντικό κόστος για την πραγματική οικονομία μέσα σε αυτό το πλαίσιο γενικότερα ένα φυσικό ερώτημα είναι αν η νομισματική πολιτική θα πρέπει να χρησιμοποιείται ενεργά ώστε να αναχαιτιστεί τέτοιου είδους φαινόμενο φούσκας. Μια απάντηση που καλούμε leaning against the wind και χάρη στην ε, νομισματική πολιτική και στρατηγική μας επικεντρωνόμαστε σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, ε, εκτιμώντας ε, τις επιπτώσεις στην σταθερότητα των τιμών. Τούτων λεχθέντων πρώτα, Ας είναι σαφές ότι οι αλλαγές στην πολιτική των επιτοκίων δεν είναι το πρώτο μέσο για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ασύμετρες σχέσεις. Πρέπει μόνο υπό έκτακτο καθεστώς να εξετάζονται όταν υπάρχει για παράδειγμα πρόβλημα όσον αφορά την διασφάλιση του περιβάλλοντος σταθερότητος τιμών στη ζώνη ευρώ συνολικά. Καθώς ε, βλέπουμε ότι ε, μπορεί να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ε, ανισορροπίες, θα πρέπει να υπάρξουν δυνατότητες ευθυγραμμίσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Για να αποφύγουμε την αύξηση των κινδύνων στον χρηματοοικονομικό τομέα ή στον τομέα στέγασης, οι εθνικές αρχές έχουν τα ενδεδειγμένα μέτρα από πλευράς φορολογίας και εποπτείας στη διάθεσή τους ώστε να δρουν έγκαιρα. Ας στραφώ τώρα στο δεύτερο ε, θέμα το οποίο επιλέξατε την δημιουργία ενός ε, ενιαίου μηχανισμού επίλυσης ε, κρίσεων, προβλημάτων. Αυτό είναι το δεύτερο, ο δεύτερος πυλώνας της Χρηματοοικονομικής Ένωσης αναγκαίο συμπλήρωμα στον πρώτο πυλώνα και στον, ε, στη διαδικασία υποπτία. Ο ενιαίος μηχανισμός αυτός θα πρέπει να επικεντρώνεται σε μία αρχή επίλυσης ε, προβλημάτων με ένα ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο θα δρά ως μέσο για αυτή την αρχή. Καλωσορίζουμε την δήλωση του Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου ότι κατά τη διάρκεια του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση για ένα τέτοιου είδους μηχανισμό ώστε τα κράτη-μέλη τα οποία θα συμμετέχουν στον ενιαίο αυτό εποπτικό μηχανισμό να μπορούν να δρουν από κοινού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη χρονική στιγμή για την λειτουργία αυτού του ενιαίου μηχανισμού με το ότι δηλαδή θα, θα απαιτηθεί η ενιαία εποπτεία που θα είναι έργο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό καλωσορίζουμε το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση στους συνομοθέτες να εξετάσουν αυτή την νομική πρότα, νομοθετική πρόταση ως πρώτη προτεραιότητα με την πρόθεση να υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κοινοβουλευτικού κύκλου της, ε, του, της Ευρωβουλής. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι λόγοι για έναν τέτοιο ενιαίο μηχανισμό με μια ενιαία εποπτική αρχή και αρχή επίλυσης προβλημάτων στον πυρήνα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μια τέτοια αρχή θα μπορεί έγκαιρα να δρά επικεντρωνόμενη στην ευρωπαϊκή διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κατάσταση όπου διασυνοριακά θα χρειαζόταν μια τέτοιου είδους δράση επίλυσης προβλημάτων, η ενιαία αυτή αρχή θα απέφευγε τον, την εστίαση σε εθνικό επίπεδο και θα ακολουθούσε την βέλτιστη στρατηγική ε, μειώνοντας τριβές και προβλήματα συντονισμού. Ο δεύτερος λόγος θα είναι ότι η ενιαία αυτή αρχή θα ακολουθεί αξιόπιστα μια πολιτική αντιμετώπισης προβλημάτων αξιολογώντας διασυνοριακά τις επιπτώσεις και τους συστημικούς κινδύνους και διασφαλίζοντας ότι θα είναι ε, στα χέρια του ιδιωτικού τομέα μια τέτοια δράση. Αυτό θα μείωνε το κόστος χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση των φορολογουμένων ο τρίτος λόγος είναι ότι μια τέτοια ενιαία αρχή είναι αναγκαίο συμπλήρωμα στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα δίνει έγκαιρα μια σωστή αξιολόγηση για την ανάγκη δράσης και επίλυσης προβλημάτων, ενώ η ενιαία αυτή αρχή θα διασφαλίζει την άμεση λήψη δράσεων όσον αφορά την ανάγκη σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και αυτό θα οδηγεί στο να παραμένει η, ε, ο συντονισμός και η εποπτεία στο ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ η, δραστηριοποίηση θα μπορεί να εξακολουθεί να παραμένει εθνική. Ο τέταρτος λόγος είναι το ότι θα βοηθήσει να διαραγεί ο φαύλος κύκλος αυτός ο μηχανισμός. Θα πρέπει αυτή η ενιαία αρχή να είναι ισχυρή και αποτελεσματική. Αυτό απαιτεί τρεις όρους για να επιτευχθεί. Πρώτον, αυτή η αρχή θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της ένα αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας. Ένα πλαίσιο λειτουργίας που θα δίνει εργαλεία και μέσα για να δραστηριοποιηθεί αυτή η αρχή αποτελεσματικά. Θα πρέπει έτσι σε σχέση με αυτή την οδηγία να θεωρήσουμε ότι αυτό έχει ρόλο κλειδιού. Η υιοθέτηση της οδηγίας ή δυνατόν κατά τον Ιούνιο είναι κατεπηγόντως αναγκαία προϋπόθεση ως βήμα για να διασφαλίσουμε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεύτερον, η ενιαία αυτή αρχή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην χρηματοδότηση επιλύσεως αυτών των προβλημάτων. Θα πρέπει να έχει λοιπόν ένα ευρωπαϊκό ταμείο στη διάθεσή της, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα με μια αξιολόγηση κινδύνων εξ άντε, εισφορών εξ Έτσι λοιπόν ο μηχανισμός αυτός θα υποστηρίζεται και από την αναγκαία δημόσια ή κρατική υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να συμπληρωθούν τα έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι ε, αμερόληπτη και ουδέτερη μεσοπρόθεσμα στη δράση της αυτή η αρχή. Τρίτον, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να είναι αποτελεσματική στη δράση της και να έχει ένα ισχυρό πλαίσιο λογοδοσίας με αποτελεσματική δικαστική προστασία σε σχέση με κάποιες αποφάσεις που μπορούσαν να ληφθούν εξ post, εκ των υστέρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή αξιολογεί τις ε, εναλλακτικέ δυνατότητες για την κατοχήρωση των δράσεων αυτής της, ε, αρχής. Προσβλέπω στις ε, προτάσεις αυτές ε, που θα διασφαλίζουν αυτές τις τρεις αναγκαίες προϋποθέσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας τώρα να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you, Mario, and, and thank you for your... Ευχαριστούμε Μάριο και σας ευχαριστούμε και για κάποια σχόλια για την νομοθεσία που πρέπει να υλοποιηθεί και να επιτευχθεί είναι πολύ θετικό σε σχέση με το Συμβούλιο όταν γίνονται κάποια πράγματα. Για να γίνουν κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχει και μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την ενιαία αρχή επίλυσης ε, δεν, δεν, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια δυνατότητα αν ε, δεν λειτουργήσουν τα πράγματα μέχρι τις ε, θερινές διακοπές να τα καταφέρουμε με άλλο τρόπο. Και γι' αυτό πραγματικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα δεδομένα και εδώ βρίσκεται ακριβώς ε, ε, το ζήτημα. Επίσης ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα σε σχέση με την ενιαία, τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και γι' αυτό ζητήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προσέλθει και να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Και προσβλέπουμε στο να προσέλθει κάποιος στις 26 Φεβρουαρίου σε σχέση με αυτά και να δώσει κάποιες διευκρινήσεις, γιατί πρέπει να τα εξετάσουμε σε βάθος και επαρκώς όλα αυτά. Είμαστε συνομοθέτες και πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο μας με τον καλύτερο τρόπο. Περνώντας λοιπόν τώρα στον γύρο ερωτήσεων-απαντήσεων. Ο Ζων Πολ Γκοζές πρώτος για το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας δώσω Συγγνώμη για εξ μέρους των ε, μελών που ε, καταλαμβάνουν, φτάνουν μάλλον ε, καθυστερημένα γιατί υπήρχε μια συνεδρία με τον κύριο Μπαρόσο και τον κύριο Βαν Ρόμποϊ και έπρεπε και εκεί να ακουστούν και οι θέσει των βασικών ε, κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα που αναφέρετε κι εσείς σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη και την ανάκτηση της εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές ε, που σήμερα είναι αρκετά ελλειπής. Και υπήρξε αυτό το διαζύγιο των εισαγωγικών ε, ε, στο μυαλό των πολιτών και τώρα πλέον ανακάμπτει. βεβαίως υπήρχε και αυτή η έλλειψη βελτίωση στην πραγματική οικονομία. Και αυτό το βλέπουμε με το κλείσμα των εργαστασίων, τις απολύσεις και την ε, ε, αποχώρηση των επενδύσεων. Επομένω, σημαντικά τα όσα είπατε, αλλά θα ήθελα να μας δώσετε και την εκτίμησή σας σε ό,τι αφορά αυτή την κατάσταση. Αν μπορείτε λίγο πιο συγκεκριμένα. Και για τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ευνοήσουν ε, αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ναι, συμφωνώ. Έχουμε κάνει πολλά από πλευρά χρηματοδότηση για να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζε θα έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα και πολλέ από τι ενέργειε που έχουμε αναλάβει τον τελευταίο χρόνο έχουν ε, θετικά αποτελέσματα, έχουν πετύχει δηλαδή αυτό το στόχο. Αποφύγαμε ε, την ευρεία τραπεζική κρίση, ιδίω ε, στο πρώτο εξάμεινο του 2012. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους οι τράπεζες δεν ε, δανείζουν στην πραγματική οικονομία. Η έλλειψη ε, πόρων, η έλλειψη κεφαλαίου και τρίτον η αποφυγή κινδύνων. Εμείς έχουμε επιλύσει το πρώτο. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την, το δεύτερο, τη δεύτερη αιτία, την έλλειψη κεφαλαίου και σίγουρα όχι την τρίτη πηγή. Πολύ συχνά μας ε, ρωτούν γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνουν άλλε κεντρικέ ε, τράπεζες, ότι η χρηματοδότηση δηλαδή θα πρέπει να εξαρτάται και να ως προϋπόθεση να έχει την, το νέο δανεισμό. Σε ένα βαθμό το κάναμε. Είπαμε στι τράπεζες ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δανειοδότηση προς τους πελάτες ως ε, ε, collateral για να λάβουν περαιτέρω ως εγγύηση, για να λάβουν περαιτέρω χρηματοδότηση από την ε, Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει όμως κι άλλος λόγος που δεν ενισχύονται αυτές οι τραπεζικές ροές και είναι η έλλειψη ζήτησης. Αναμφίβολα, με την... με τις δυσμενείς επιπτώσεις στον επιχειρηματικό κύκλο δεν αυξάνεται η ζήτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Πρέπει να περιμένουμε να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους οι τράπεζες για να δώσουν και δάνεια. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως η ολοκλήρωση της ε, ε, τραπεζικής ε, ένωσης για να διαμορφώσουμε αυτό το συνολικό πλαίσιο, όμως βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να περιμένουμε, ούτω ώστε η κοινή μα ε, θέση θα βρει τον δρόμο να φτάσει στην ε, πραγματική οικονομία. Εν τω μεταξύ, είχαμε ένα εξαιρετικά δύναμο τέταρτο τρίμηνο. όπω είπα όμω και στην εισαγωγή μου, όλοι οι δείκτες μελετών δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή έχει σταθεροποιηθεί στα χαμηλά αυτά επίπεδα. Πρέπει τώρα λοιπόν να περιμένουμε για αυτό το ε, δυναμικό κίνητρο από αυτό το χαμηλό επίπεδο επιτοκίων και παρεμπιπτόντως συνεχίζουμε ε, ακριβώς ε, σε αυτή την οδό και αυτά τα overnight interest ε, rates είναι κοντά στο 0%. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να φτάσουν αυτά στην οικονομία. Μέτρα για την ε, αύξηση των κεφαλαίων ε, των τραπεζών δεν αφορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά τις εθνικές αρχές και κυβερνήσεις. Τούτου λεχθέντος θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τρόπους και μέσα Βελτίωση αυτή τη μεταφορά τη νομισματικής μα πολιτική στην πραγματική οικονομία. Γιατί αναμφίβολα αυτή είναι η παριθμόν ένα πρόκληση για μα. Και δεν θέλω να υποτιμήσω αυτή τη τυχή σε κανένα επίπεδο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ευχαριστώ. S&D Φεραίρα, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε ανάμεσά μας, κύριε Ντράγκη. Για αυτές τις νέες δυνατότητες σε σχέση με τα, τις πιστώσεις, τα δάνεια, τραπεζικά δάνεια και σε σχέση με τις, ε, τα προβλήματα της κρατικής υπερχρέωσης ε, και καθώς ε, αφορά επίσης και την επίλυση των προβλημάτων τραπεζών. Αλλά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένα από αυτά. Είναι η ύφεση στη ζώνη ευρώ, ιδιαίτερα ύφεση στη ζώνη ευρώ ακριβώς. Αυτή τη στιγμή σε μια χώρα που σε σχέση με τις συστάσεις ε, της Τρόικας ε, που ακολουθήθηκαν αναμενόταν ότι θα είχαμε μια ύφεση και 2,8 ε, να έχουμε 3 και παραπάνω. Τώρα αναμέναμε ότι ε, θα υπήρχε αυτή η κατάσταση και τώρα έχουμε πρόβλημα πάρα πολύ έντονο. Μας ε, δίνει ένα περιθώριο προσαρμογών το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει σε μεγαλύτερο χρόνο, με σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και με λιγότερο βία μέτρα. Θα λάβει υπόψη η Ευρώπη αυτά τα θέματα όταν από πλευρά της Τρόικας θα αναλυθούν οι επιτυχίες, οι αποτυχίες αυτών των δράσεων σε σχέση με τις συγκεκριμένες χώρες. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω ευθύ εξ αρχή για αυτό το θέμα, επειδή όπω είπα είναι η κυριότερη πρόκληση αυτό για μα. Τι μπορούμε, να, κάνουμε. δηλαδή. Τι μπορούμε να κάνουμε. Θα ήθελα να πω με πολύ εμφατικό τρόπο ότι ξέρουμε πολύ καλά τι συνθήκε μέσα στι οποίε. Ε, πολλές από τις χώρες Ευρωζώνης ε, ζουν και λειτουργούν. Η δημοσιονομική εξυγίανση, ειδικά για χώρες με υψηλό χρέος, είναι αναπόφευκτη. Παράλληλα, σωστό είναι ότι βραχυπρόθεσμα θα υπάρξει μια συρρήκνωση. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε να αναβάλουμε τόσο ή αν μπορούμε να αναβάλουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση ή αν θα τη μετριάσουμε. Το θέμα είναι πώς θα μετριάσουμε τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής εξυγίανσης που θα κάνουμε. Όχι να μειώσουμε την ίδια τη δημοσιονομική εξυγίανση. Πώς πετυχαίνουμε το μετριάσμα των επιπτώσεών της. Αν σχεδιάσουμε σωστά την δημοσιονομική εξυγίανση, και να βασίζεται περισσότερο στις, ε, στη μείωση των δαπανών και όχι στην αύξηση των φόρων. Θα πω κάτι που δεν είναι οικουμενική αλήθεια, αλλά για τις χώρες Ευρωζώνης οι, φόροι είναι ήδη πολύ ψηλοί. Το δεύτερο είναι η εφαρμογή, η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και στην αγορά προϊόντων. Και το είδαμε σε μια-δυο χώρε. Γιατί είδαμε ότι αν γίνει αυτό, θα δούμε ότι αυξάνονται οι εξαγωγέ. Και επομένω έχουμε τουλάχιστον μια συνιστόσα του ΑΕΠ που δεν κατεβαίνει. Έχετε την κατανάλωση που κατεβαίνει, έχετε τι επενδύσει που, κατεβαίνουν, που πέφτουν ε, βραχυπρόθεσμα, αλλά τουλάχιστον ε, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κάτι αυξάνεται και έτσι μετριάζεται τις α, ε, βραχυπρόθεσμα τις επιπτώσεις αυτές της συρρήκνωσης από την εφαρμογή Τη δημοσιονομική εξυγίανση. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Η αξιοπιστία των σχεδίων των χωρών αυτών. Αν έχουν μεσοπρόθεσμα, λεπτομερή, δημοσιονομική σχέδια, δημοσιονομικά σχέδια και προγραμματισμό, αυτό καθησυχάζει τις αγορές. Αυτά τα ε, προγράμματα όμως, τα, τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Και όσο υψηλότερη βέβαια είναι η λεπτομέρεια σε αυτά τα προγράμματα, τόσο υψηλότερο είναι και το πολιτικό κόστο. Αλλά όμω το όφελο είναι μεγαλύτερο γιατί υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Σημαίνει ότι έχουμε χαμηλότερα επιτόκια κτλ. Και, και χαμηλότερε τιμέ βέβαια. Θε να επανέλθει κυρία Φερέιρα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν είναι το θέμα εδώ η προσαρμογή είναι η διάρκεια της προσαρμογής και η διάσταση της προσαρμογής γιατί 70% ε, των αγορών σε σχέση με τις εξαγωγές βρίσκονται σε ύφεση οι χώρες της ζώνης ευρώ και οι χώρες της Ευρώπης και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, οικονομετρικά όσα προτείνονται θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια προσαρμογή και που θα λαμβάνει υπόψη αυτά τα προβλήματα για τις χώρες και γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να πείτε ότι συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη χώρα, στην κάθε χώρα. Δεν έχουμε ένα γενικό πλαίσιο που κάνει για όλους. Παράλληλα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ταχύτητα και ο ρυθμός της δημοσιονομικής εξυγίανσης εξαρτάται επίσης από το επίπεδο του χρέους, από το αρχικό επίπεδο του χρέους. Άρα από τις ε, συνθήκες Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε στι συνθήκε. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να μετριάσουμε δηλαδή, τη δημοσιονομική εξυγίανση, αυτό εννοείται. Όχι, εμεί δεν, εννοούμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μετριασμό των επιπτώσεων τη εξυγίανση αυτή. Αλλά η αποδυνάμωση τη εξυγίανση αυτή θα οδηγούσε στην απώλεια κάποιων από τα ωφέλη. Ε, Ούτω ή άλλω έχουν γίνει θυσίε. Άρα θα ήταν κρίμα να χάσουμε τα ωφέλη. Και επομένω πραγματικά ε, είναι μια λεπτή ισορροπία. Φιλελεύθερη. Κύριε Πρόεδρε, έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, αυτό ο, ο ε, πόλεμο, ο συνολματικό πόλεμο και δεύτερον η Κύπρο. Καταστήστε σαφέ τι εισαγωγικέ σα ε, ε, παρατηρήσει ότι δεν ε, πρόκειται για συγκεκριμένο στόχο εδώ πέρα, όμως αυτή δεν είναι πολιτική όλων των ε, ε, μελών του G20. Η Ιαπωνία και άλλες χώρες ε, θέλουν, έχουν μια ενεργή πολιτική για την αλλαγή των συναλλαγματικών ιστομιών και αυτό έχει φανεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και με την παρέμβαση της Ελβετίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν αλλαγές λοιπόν στην ατζέντα του G20, τα αποτελέσματα ε, όμως ήταν αρνητικά, ανέβηκε 2% στην Ιαπωνία ε, το χρηματιστήριο, γιατί είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πλέον. Επομένω, ε, ποια είναι η εκτίμηση εδώ. Δεύτερον, ε, για την Κύπρο. Ε, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, από όλα τα κόμματα κατέστη σαφές ότι δεν θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε ένα τέτοιο πακέτο στήριξη της Κύπρου εκτός και αν η Κύπρος ε, υιοθετήσει κάποιε πολύ σημαντικέ ε, αποφάσει ε, κατά του ξεπλήματος βρωμικού χρήματος της καταπολέμησης του tax dumping, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις Όσοι έχουν αποφεληθεί από το ξέπλυμα χρήματος ε, συμμετείχαν στην όλη διαδικασία και ξέρετε σε ποιους αναφέρομαι και ε, εισήγαγαν αυτόν τον, ε, κόστο, τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Κατά τη δική σας εκτίμηση λοιπόν, σε τι βαθμό θα μπορέσει η κυπριακή κυβέρνηση να τηρήσει αυτές τις προσδοκίες. Ευχαριστώ. Για το πρώτο ζήτημα, για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι ισοτομίες αντικατοπτρίζουν την ουσία. Αν εξετάσουμε την ονομαστική και πραγματική επίπτωση ε, της ισοτομίας ε, του ευρώ, βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές είμαστε περίπου στα μακροπρόθεσμες μέσες τιμές. Αυτό καθορίστηκε από ε, το στην τελευταία συνάντηση G20. Ε, βεβαίως και οι ισοτιμίες δεν είναι το στόχος πολιτικής και το επαναλαμβάνω. Όμως οι ισοτιμίες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών. Και πρέπει να εκτιμήσουμε στις επόμενες ε, ε, μελλοντικέ αν αυτές οι ισοτομίες έχουν αντίκτυπο στο προφίλ μας. Γιατί μέσω των ε, μέσω της σταθερότητας των τιμών αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα. Για τα υπόλοιπα μπορώ μόνο να πω ότι η ανακοίνωση του G20 δεν είναι και τόσο απογοητευτική κατά τη γνώμη μου. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να κινηθούμε πιο γρήγορα προς ε, καλύτερα συστήματα ισοτιμίας και ευελιξίας των ισοτιμιών για αποφευθούν ε, οι μεγάλες ενωσορροπίες και όπως και να έχει θα συνεργαστούμε πιο στενά για να αναπτυχθούμε από κοινού. Δεν θέλω να συνεχίσω γιατί ουσιαστικά είναι η ε, καθιερωμένη διατύπωση που χρησιμοποιείται. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ένα άλλο στοιχείο. Οι περισσότερες από τις κινήσεις ε, ισοτιμιών που έχουμε παρατηρήσει δεν είχαν ρητό στόχο ήταν ε, απόρρια ε, μακροπρόθεσμων μακροοικονομικών πολιτικών με στόχο την ενίσχυση της αγοράς. Έτσι, δεν μπορούμε ακριβώ να πούμε και το θεωρώ και υπερβολικό αν θέλετε οτιδήποτε αναφέρεται σε ε, πόλεμο ισοτιμιών και το καθεξής. Ουσιαστικά το G20 καλεί όλα τα μέλη σε πολύ ισχυρή λεκτική πειθαρχία. Για την Κύπρο να σα πω ποια είναι η θέση. Ε, χαιρετίζουμε τη δέσμευση της κυπριακής ε, κυβέρνηση, ε, να καταρτήσει μνημόνιο κατανόησης και εκτιμούμε και τις προσπάθειες υιοθέτηση των πρώτων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί. Τώρα, μετά τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, είναι πολύ σημαντικό να συμφωνηθεί το πρόγραμμα. Η δήλωση του Eurogroup λέει ότι θα υπάρξει πρόγραμμα και πρέπει να συμφωνηθεί. Είναι Θεμελιώδους σημασία λοιπόν να υπάρξει ε, πραγματική δέσμευση από πλευρά κυβέρνηση μετά τι εκλογέ. Πρέπει να βρούμε επίση τρόπου ε, διασφάλιση τη βιωσιμότητα αυτού του, του προγράμματο. Δεν θέλω να προδικάσω τι συζητήσει ε, που θα λάβουν χώρα για να δούμε πώς ακριβώς θα υπάρξει αυτή η βιωσιμότητα. Όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε δύο πλευρές. Αφενός θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος θα έχει αυτή την βιωσιμότητα. Αφετέρου πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουμε δημοσιονομική αστάθεια. Πρέπει λοιπόν και οι δύο αυτές πτυχές ε, να υπάρχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μετά, σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση, διαφάνεια και εποπτεία του, τραπεζι... του χρηματοοικονομικού τομέα, θα πρέπει να ενισχυθούν. Ε, σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, τη δανειοδότηση ε, και τη δημοσίευση, όλα αυτά θα αναθεωρηθούν μέχρι το 2013 και για να απαντήσω στο τελευταίο τμήμα της ερώτησής σας, η τελική εκδοχή του προγράμματος ε, προσαρμογής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και στενή ε, ε, εποπτεία των πλαισίων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του ξεπλήματο χρήματο. Δηλαδή, όχι μόνο λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει τέτοια νομοθεσία, αλλά και να εφαρμοστεί. Εμεί θα πρέπει να διασφαλίσουμε την εφαρμογή τη. Αυτά είναι ακριβώς και από το έγγραφο το οποίο ε, είναι ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα και σε σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπέζα. Σας ευχαριστώ. Εσείς ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι προφανές. Μικρόφωνο. Ναι. εδώ θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική εργαλειοθήκη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με βάση αυτές τις σημαντικές αποφάσεις. Και πιο σημαντικό είναι το ότι αναγνωρίζουμε την σύνδεση σε σχέση με τις ε, τράπεζες και που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και ο ενιαίος εποπτικός ε, μηχανισμός, ε, το πρώτο δηλαδή σκέλος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης που θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί και να υπάρχει η δυνατότητα δραστηριοποίησης της Ευρωζώνης και των τραπεζών της ε, και να αποκατασταθεί η λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς σε σχέση με αυτές τις αγορές ε, όχι μόνο των χωρών ε, της Ευρωζώνης αλλά και ευρύτερα. Σημαντικό αυτό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με σωστό τρόπο. Ήδη περιγράψατε επαρκώς αυτά και σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας για τον μηχανισμό επίλυσης ε, ε, των προβλημάτων και για κάποια πιθανή ε, καθυστέρηση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να υπάρχει η πρόσβαση σε σχέση με τις τράπεζες σε αυτό το μέσο με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις αλλά για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης δεν θα μπορεί να προβληθεί βλέπετε, κάτι τέτοιο, εκτό από κάποιο κατεπίγοντα, ε, κάποια κατεπίουσα περίπτωση. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε αυτή την περίπτωση ακριβώς, τι θα μπορούσε να γίνει σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, δηλαδή δύο διαφορετικών ε, ομάδων χωρών ε, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι ε, το SSM στρεβλώνει την λειτουργία της ε, ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Και μάλιστα θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί την λειτουργία του SSM ως ένα μέρος, ε, ως ένα συμπλήρωμα του EBA, στις δράσεις του EBA. Το SSM λοιπόν θα έπρεπε να μπορεί να βοηθήσει το EBA για να λειτουργήσουν τα πράγματα σωστά και με την λειτουργία βέλτιστων πρακτικών με ενιαίο τρόπο σε σχέση με τις ε, ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να συνεισφέρει και το EBA από πλευρά ε, ε, αυτών των δράσεων. Τώρα για το ESM και το δυναμικό το οποίο υπάρχει για την δυνατότητα αναχρηματοδότησης άμεσα των τραπεζών. Ένα πράγμα πρέπει να θυμόμαστε ότι και οι χώρες εκτός Ευρωζώνης μπορούν να ενταχθούν ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και έτσι θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες ε, για τις ε, δράσεις του ESM για την άμεση κεφαλαιοποίηση, ανακεφαλαιοποίηση όταν αυτό το μέσο θα μπορεί να λειτουργεί πλήρως. Ευχαριστώ. Εσείς θέλατε να επανέλθετε με επερώτηση, παρακαλώ. Μπορείτε να θέσετε επερώτηση πολύ σύντομα γιατί πρέπει να το κατανοήσουμε σωστά. Η απόφαση ε, της ε, ε, Συνόδου Κορυφής ήταν ότι μόνο οι χώρες της Ευρωζώνης θα μπορούν να κεφαλοποιούνται, να επαναχρηματοδοτούνται από το ESM. E Τώρα, για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης που ε, σε σχέση με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό που θα μπορούσαν να έχουν μια δυνατότητα χρηματοδότησης από το ESM. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετηθήκατε. Εγώ είπα ότι χώρες εκτός ζώνης ευρώ θα μπορούσαν να ενταχθούν στο ESM και στο SSM και τότε θα ε, υπόκεινται στον ενιαίο εποπτικό τραπεζικό μηχανισμό και έτσι θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες, ε, δυνάμει επιλέξιμες για την κεφαλαιοποίηση αυτή υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ESM. Δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να ε, διαχωρίσουμε ή να διχάσουμε, να κατακαιρματίσουμε την ενιαία εσωτερική αγορά θα έπρεπε να μπορούμε να δούμε μια συνεισφορά από πλευρά μα για την βέλτιστη λειτουργία, ε, τη ενιαία εσωτερική αγορά με αυτά τα μέτρα. Ικανοποιήστε με την απάντηση αυτή. Οι νομικές μου γνώσεις δεν επαρκούν ε, ίσως, αλλά καθότι είχε συζητηθεί και έκθεση σχετικά για αυτό το θέμα, υπάρχουν νομικά εμπόδια και προσκόμματα από ό,τι φαίνεται για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης να ενταχθούν στο ESM. Αυτό ήταν η ερώτηση, αυτό ήταν ο λόγος της ερώτησής μου. Σε αυτό το ε, σημείο θα ήθελα να πω ότι αυτή ήταν η δική μου πεποίθηση, αλλά ίσως ε, εδώ υπάρχουν και ε, άλλες απόψεις που μπορούν να διαφοροποιήσουν αυτή την άποψη. Τώρα για το πώς θα μπορέσει να ε, τετραγωνιστεί ο κύκλος ε, είναι ζήτημα αυτό. Περνάμε στην ενωτική αριστερά παρακαλώ στην Όχι, συγγνώμη, περνάμε στους πράσινους ε, πρώτα. Συγγνώμη Φιλίπ, δεν σας είδα πιο πριν, εσείς. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε ακόμα μια φορά όπως πάντα. Παρότι σας κέρδισε η πολιτική, να σας επιστήσω την προσοχή στα εξής. Είπατε ότι η φόρη είναι υψηλή στην Ευρώπη. Είναι πολιτική δήλωση αυτή. Ε, θέλετε να πείτε μήπως ότι είναι συγκριτικά υψηλότερες, ε, υψηλότεροι φόροι ε, στην Ευρώπη. Γιατί το άλλο είναι πραγματικά πολιτική δήλωση και δεν ξέρω αν εμπίπτει στην εντολή σας να λέτε κάτι τέτοιο. Επίσης, είπατε ότι η επίπτωση της δημοσιονομικής περιχαράκωσης είναι αρνητική βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή θα πρέπει να μετριάσουμε τις επιπτώσεις, αλλά όχι την εξυγίανση. Επίσης για τις τράπεζες είπατε ότι υπάρχει αρνητική επίπτωση στην απομόχλευση και θα πρέπει να επιβραδύνουμε την απομόχλευση. Αυτά όταν κάνετε τις παρατηρήσεις σας ε, στα τέλη του 12 για ε, το θέμα της ρευστότητας. Τώρα, Μιλήσαμε για την εποπτεία του, της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Για την ε, Ιρλανδική αναχρηματοδότηση. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό που έγινε για την Ιρλανδία έγινε χωρίς την συνένεση της ε, ΕΚΤΑ. Θα, ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα για την Ιρλανδία. Αν θέλετε να πείτε δηλαδή κάποια πράγματα. Μπορείς περιπτώσει θα τα άκουγα με ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια. Δεν θα σχολιάσω αν η δήλωσή μου ήταν πολιτική ή όχι. Θεωρώ ότι είναι γεγονός. Εσείς μπορείτε να το θεωρήσετε ε, πολιτική δήλωση ή όχι. Το 3% για το Google είναι υψηλό, λέει ο μιλητής. Η ουσία ήταν αυτή πάντως που είπα ότι υψηλή είναι η φόρη. Τώρα για την απομόχλευση των τραπεζών. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να επιβραδύνουμε την απομόχλευση των τραπεζών. Δεν είπα αυτό. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε, και νομίζω το πέτυχε η ΕΚΤ πέρυσι, είναι να αποφύγουμε μία άτακτη απομόχλευση. Να σας δώσω ένα θετικό παράδειγμα του τι συνέβη ας πούμε στην Ισπανία. Με τη δημιουργία αυτής της εταιρείας ε, οι τράπεζες μπορούσαν να μεταφέρουν ε, σε μετριοπαθείς συντηρητικές τιμές στοιχεία του ενεργητικού σε αυτή την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που αλλιώς θα πουλιόταν με τρόπο άτακτο. Αυτές οι πωλήσει είναι αποσταθεροποιητικές και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και άλλες αυτοεπιρούμενες καταστροφές. Εγώ δεν είπα ότι θα πρέπει να επιβραδύνουμε την απομόχλευση, κάτι που χρειαζόμαστε. Γιατί αν δεν κάνουν την δική του σωστή απομόχλευση, δεν θα υπάρξει, θα ρυθμίσουμε το θέμα της ε, πίστοσης. Και αυτή είναι η βασική μας πρόκληση. Θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη πίστοση στην ΕΠΗ για την Ιρλανδική κατάσταση. Το σημείωσα αυτό που είπατε. Είναι μια συναλλαγή μεταξύ της Ιρλανδικής κυβέρνησης και της ε, Κεντρικής της Τράπεζας. Το Δουσού δεν χρειάστηκε να αποφανθεί. Θα το κάνει στα πλαίσια της ετήσιας αξιολόγησης για την ε, οικονομική κατάσταση στις, για τις ε, κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Δηλαδή, θα γίνει μια αξιολόγηση με βάση το άρθρο 113. Αλλά όχι σε αυτή τη φάση. Είχαμε μια, ε, ένα μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης, δανεισμού στην ε, ε, Ιρλανδία. Επί πολλά χρόνια. Αλλά αυτό εξαφανίστηκε τώρα και υπάρχουν κάποια ομόλογα που μπορούν να απολυθούν και που η Κεντρική Τράπεζα θα, μπορούσε, θα τα πουλήσει το συντομότερο ε, δυνατό. Δεν θέλω να αποφανθώ, αλλά οι εξελίξεις, κάποιες εξελίξεις, ε, νομίζω ότι σε όλες τις ήταν θετικές. Κάτι σημαντικό για το μέλλον και ίσως απαντάω έτσι και σε άλλες ερωτήσεις. Θα είναι η πολιτική διάθεση αυτών των ομολόγων από την Κεντρική Τράπεζα. Αλλά το Δουσού για να αξιολογήσει αυτή την κατάσταση θα την κάνει ε, σε τακτά διαστήματα, την κάνει στα πλαίσια δηλαδή του κάθε έτους. Και τώρα πάμε στην ΚΟΕ. Μαρίσα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ κύριε Ντράγκη. Κάνατε λόγο για τα χαμηλά ποσοστά και για το επιτόκια και για το ε, χαμηλά επιτόκια που όμως ε, πολλές φορές ε, δεν δίνουν εκείνο το αποτέλεσμα το οποίο επιθυμούμε. Και βλέπουμε μια ύφεση ταυτόχρονα και συμφωνώ με αυτό. Και έχουμε και σε άλλες χώρες και τη ζώνη ευρώ και στη Γερμανία παρόμοια προβλήματα. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε το τι μπορεί να γίνει σε σχέση με μια πολιτική για την ανάπτυξη που να δώσει δυνατότητα ανάπτυξης. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς βλέπετε εσείς μια τέτοια συμπερίληψη μιας πολιτικής ε, δημοσιονομικής για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για να αντιμετωπιστεί η ύφεση, μια και δεν δίνουν το ευταίο αποτέλεσμα τα χαμηλά επιτόκια. Και σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα εδώ για το πρόβλημα του ότι ε, δεν υπάρχει ρευστότητα στην οικονομία. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που παρουσιάστηκαν. Εδώ αναφέρθηκαν τρεις λόγοι για αυτή την κατάσταση. Έλλειψη κεφαλαίου, έλλειψη ρευστότητας, ε, κίνδυνοι που υφίστανται. Και εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε στην έλλειψη της ρευστότητας. Υπάρχει και ένας τέταρτος όρος, οι όροι και οι προϋποθέσεις ε, είναι θεμητό να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε σχέση με τα δάνεια στο επίπεδο των ε, χωρών μας χωρίς όρους και προϋποθέσεις για τις τράπεζες για τέτοιου είδους δανειοδοτικές πράξεις. Θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη πολιτική. Εφόσον δεν θα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις με συγκεκριμένους στόχους, τότε τι θα κάνουμε. Θα ε, λειτουργούμε χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτά είναι που πρέπει να λάβουμε υπόψη σε σχέση με αυτό το τέταρτο στοιχείο που ανέφερα, αν μπορείτε να το καλύψετε. Ευχαριστώ. Well, Όπως προανέφερα, κάναμε πολλά ήδη σε σχέση με την αύξηση της ρευστότητας ε, για το χρηματοοικονομικό σύστημα και βλέπουμε ήδη τα πρώτα ωφέλη ήδη. Δεν θέλω να το αμελήσουμε αυτό. Είδαμε για παράδειγμα ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις επανέρχονται πάλι στις αγορές και μπορούν ε, να χρηματοδοτηθούν με την έκδοση ε, ομολόγων, εταιρικών ομολόγων. Όμως, ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, το πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα και που πλήττει περισσότερο την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 75% περίπου της απασχόλησης στη ζώνη ευρώ και οι περισσότερες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η πρόκληση λοιπόν που ανέφερα στην αρχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι αυτή ακριβώς. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια κατάσταση μέσω της οποίας η ρευστότητα που ε, δίνουμε στο σύστημα θα μπορέσει να περάσει από το τραπεζικό σύστημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό εξακολουθεί να είναι πρόκληση και εξακολουθούμε να προβληματιζόμαστε σε σχέση με αυτό. Βλέποντας τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο όμως, δεν θεωρούμε σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία ότι κάναμε λιγότερα εμείς από ό,τι άλλοι μέσα στο πλαίσιο των συγκεκριμένων θεσμών που έχουμε και που λειτουργούν στη ζώνη ευρώ. Παράδειγμα, έχουμε τράπεζες που καλύπτουν 80% για παράδειγμα αυτής της ε, χρηματοδότησης. Δεν είμαστε σε μια θέση όπως άλλοι που θα μπορούσαν να αγοράσουν για παράδειγμα ε, ομόλογα της ε, ε, ευρύτερης οικονομίας και θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε σχέση με, την, με τα ωφέλη αυτά είναι μέσα από το τραπεζικό σύστημα και μέσα από αυτό το πλαίσιο πρέπει να απορρέουν. Εξακολουθούμε να προβληματιζόμαστε γι' αυτό γιατί είναι η κύρια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και πολύ άμεσα γι' αυτό δεν θεωρείτε εσείς κύριε Ντράγκη ότι ο ορισμός των όρων λειτουργίας των τραπεζών θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά πιο σωστά εφόσον τα άλλα μέτρα απέτυχαν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά σε σχέση με τα δάνεια και υπάρχει πρόσβαση απεριόριστα ώστε να μπορέσει να υπάρξει αυτή η δραστηριοποίηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα. Το να υπάρξουν όροι και προποθέσει δεν θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέτρο. Να πούμε ότι ένα συγκεκριμένο ποσό θα δίνεται για παράδειγμα στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Δεν θα ήταν μια υπόθεση εργασία αποτελεσματική αυτή. Είναι προκλητικό να μπορέσει να πει κανεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι απόλυτα σαφέ ότι με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργούν τα πράγματα αν υποχρεωθεί μια τράπεζα να δώσει τέτοια δάνεια υπό οποιασδήποτε συνθήκες σε μια εταιρεία και η εταιρεία αυτή χρεοκοπήσει, πτωχεύσει, τότε χάνει τα κεφάλαιά της αυτή η τράπεζα. Δεν θα μπορεί να διαθέτει δάνεια στις άλλες επιχειρήσεις μέσα στο πλαίσιο τη οικονομία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ποιο εύρο, σε ποιο ύψο θα θέσουμε τον πύχη με τη δημιουργία όρων και προϋποθέσεων διότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν ευθύνε, έχοντα, α το πω έτσι, επιβάλλει στο τραπεζικό σύστημα να κάνει πράγματα τα οποία συνήθω ε, δεν θα έκανε ή δεν κάνει. Με κάθε συμπάθεια για το ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση αποτελεσματικά, πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει τι ενδυνάμει αρνητικέ επιπτώσει συγκεκριμένων παρεμβάσεων στι αγορέ ε, δανείων και πιστώσεων μέσα στο σύστημά μα. Σα ευχαριστώ. Εσεί έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έχω κάποιες ερωτήσεις όπου φυσικά έχουν αναφερθεί κάποια πράγματα ήδη προηγούμενα. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως με τη Λετωνία. Τις επόμενες εβδομάδες ε, η κυβέρνηση της Λετωνίας ε, πιθανότητα θα θέσει το αίτημα να ενταχθεί στην ε, ζώνη ευρώ, στην νομισματική ένωση είχα την τιμή στο Ευρωκοινοβούλιο να παρακολουθώ αυτό το θέμα ως εισηγητής. Γι' αυτό ερώτημά μου προς εμάς, Πρόεδρε. Πώς κρίνετε εσείς ε, τα νομισματικά θέματα για τη Λετωνία και την προπαρασκευή της Λετωνίας για μια ένταξη στην Ευρωζώνη. Δεύτερη ερώτηση που αφορά τον ε, ενιαίο ε, εποπτικό τραπεζικό μηχανισμό. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία της ε, εποπτικής αυτής ε, αρχής ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και, του μηχανισμού αυτού. Και ποιος θα είναι, ποιες θα είναι οι διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με τις εθνικές τραπεζικές αρχές που με κριτικό πνεύμα αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα από το Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ το Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί διαφορετικά. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού και ποια μειονεκτήματα, μειονεκτήματα θα βλέπατε σε μια τέτοια ρύθμιση. Χωρίς μικρόφωνο. Για το πρώτο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αξιολογήσει τη σύγκληση της Λετωνίας προς τα κριτήρια που έχουν τεθεί και τους όρους και προϋποθέσεις και τις, το δυναμικό και τις ικανότητές Δεν μπορώ να προδικάσω τοποθετούμενος ε, αυτή τη στιγμή από αυτού. Για το άλλο θέμα που θέσατε, όλοι καλούμαστε και διατυπώνουμε ερωτήσει ε, σε σχέση με το πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα. Θυμόμαστε όμως κάποια πράγματα. Δεν έχει ακόμα εγκριθεί το SSM και καθότι γνωρίζετε, οι διαβουλεύσεις ε, βρίσκονται υπό εξέλιξη. Όταν θα αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός, ε, θα υποβάλει έκθεση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί στην λειτουργική εφαρμογή όλων αυτών. Και θα είναι δημόσια αυτή η έκθεση. Και σίγουρα έχουμε ξεκινήσει τις προκατακτικές μας δράσεις. Όμως δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε δεσμευτικά ή με διοικητικές δεσμευτικές αποφάσεις μέχρι ότου θα έχει εγκριθεί το νομικό κείμενο επ' αυτού. Τώρα να εκφράσει κανείς κάποια συμπεράσματα επ' αυτού είναι υπερβολικά πρόημο σε αυτό το στάδιο. Είχαμε μια μελέτη επ' αυτού, αλλά είναι μια μελέτη μεταξύ πολλών άλλων και απλώς σκιαγραφεί κάποια πράγματα και ήδη αυτά βρίσκονται ρευστό και μετεξελίσσονται ήδη. Ναι. Εντάξει, για το ΕΛΚ, θα Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε βλέπουμε ήδη θετικά μηνύματα σε σχέση με την εμπιστοσύνη όσον αφορά την αγορά, για τις ε, ε, ε, εξαγωγές, για την, την ανταγωνιστικότητα που αυξάνεται. Αλλά ακούσαμε κιόλα ότι η κυρία πρόκληση που αντιμετωπίζουν κάποιε οικονομίε, κυρίω οι οικονομίε των κρατών του Νότου, είναι οι πιστώσει και τα δάνεια στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και όπω είπε ο κύριο Γκόζε, χωρί αυτό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Και χωρί αυτά τα αποτελέσματα δεν θα έχουμε ανάκαμψη. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει συνεχίζουν να, να λειτουργούν σε σχέση με την έδρα του και για τη χρηματοδότησή του και όχι για την οικονομική του θέση. Και βλέπουμε ότι αυτό έχει ήδη επιπτώσει ε, η Financial Times σήμερα λέει ότι είναι διαφορετικό το κόστος ε, της λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων σε σχέση με την έδρα τους. Τώρα, σε σχέση με τον μηχανισμό, εποπτικό μηχανισμό, είναι το πρώτο βήμα, αλλά δεν επαρκεί πλήρως και δεν αρκεί. Και σε σχέση με την ανάλυση θα πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές δεν υπάρχει ε, ζήτηση ε, ρευστότητας. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να χρηματοδοτούνται με ε, επιτόκια θετικά και όχι με υπερβολικά επιτόκια όπως στην Ισπανία και αλλού. Να έχουμε επιτόκια τα οποία θα είναι θετικά όπως και στη Γερμανία. Αυτό θα ήταν δικαιότερο. Ευχαριστώ. Είπα πιο πριν ότι... Είπα και προηγουμένως ότι οι τράπεζες για να δανείσουν ε, εν γέννη αλλά και πιο συγκεκριμένα ε, στις μικρομεσές ε, τα ανέφερα προηγουμένως. Πράγματι υπάρχει ζήτηση. Ωστόσο, μία μελέτη της ΕΚΤ δείχνει ότι σε ορισμένες χώρες πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ διαφόρων ε, μορφών και ειδών ε, δανειολεπτών. Υπάρχουν κάποιοι που είναι υπερχρεωμένοι και δεν μπορούν να λάβουν περαιτέρω δανεισμό, άλλοι που δεν έχουν καθόλου χρέη και λαμβάνουν δανεισμό. Υπάρχει λοιπόν η ζήτηση αλλά και η σύνθεση του ισολογισμού του δανειολήπτη. Όλα αυτά μετράνε. Τώρα, σε χώρες όπου η απομόχλευση που συνεχίζεται έχει ακόμα δρόμο μπροστά της, ε, περιμένουμε ότι ο δανεισμός θα καθυστερήσει να φτάνει στην οικονομία. Γιατί οι ίδιοι οι δανειολήπτες έχουν αυτό το βάρος ε, στον ισολογισμό τους. Αυτές οι επενδύσεις πρέπει να ρευστοποιηθούν και μέχρι τότε ε, οι επενδύσεις τους απορροφούν τα κεφάλαιό τους και γι' αυτό αυτές οι επιχειρήσεις καθίστανται ακόμα λιγότερο ελκυστικές για τις τράπεζες. Γι' αυτό δεν μπορούν να βρουν ε, δανεισμό. Να περάσω τώρα στα επιτόκια, γιατί αναφερθήκατε και σε αυτό το θέμα. θεωρούμε ότι με την ανακοίνωση OMT και μετά το ε, πρόγραμμα που ακολούθησε, το οποίο σχεδίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε καθορίσει κάποιους ε, κινδύνους, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, πηγές κατακαιρματισμού. Να μην ξεχνάμε ότι ανέβηκαν τα spreads στα στεγαστικά, όχι μόνο λόγω συγκεκριμένων κινδύνων, αλλά και ε, λόγω επιπέδων ελλημάτων και προβλημάτων που δεν είχαν επιληθεί, ιδίω μετά την χρηματοοικονομική κρίση. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και πολλά σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο της, ε, του κατακαιρματισμού σε κάποιες ε, χώρες ε, οι αγορές καθορίζουν τις τιμές των ομολόγων με συγκεκριμένο τρόπο και πρέπει αυτό να αντικατοπτρίζεται και με τους κινδύνους των δανειοληπτών. Και τον δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει το κόστος του δανεισμού γιατί κάποιες τράπεζες ε, θα μπουν στον πειρασμό να αγοράσουν ομόλογα αντί να δανείσουν στον ιδιωτικό τομέα και έτσι να αυξήσουν τα κέρδη τους. Γι' αυτό η δημοσιονομική εξυγίανση και οι αδιαρθρώσεις αυτές είναι, λειτουργούν συμπληρωματικά. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να μειώσουμε τα spread στα ομόλογα και έτσι ο δανεισμός να γίνει πιο φθηνός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. και ίσως costes, esos diferentes Για αυτά τα διάφορα κόστη σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πότε νομίζετε, πώς μπορεί να επιτευχθεί να φτάσουν σε ένα όριο το οποίο θα είναι λογικό για να λειτουργήσει η ενιαία εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Όπω Όπως είπα, αυτό θα το δούμε στο δεύτερο τμήμα του χρόνου. Θα δούμε μια σταδιακή ανάκαμψη και βλέπουμε από τα δεδομένα ότι η οικονομική σταθερότητα, δραστηριότητα αυτή τη στιγμή σταθεροποιείται σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα. Έτσι, εν μέρει αυτό θα επιτευχθεί όταν ε, η πολιτική μας θέση στα νομισματικά ζητήματα που παραμένει ε, βρει τον δρόμο να φτάσει στην ε, πραγματική οικονομία. Όμως αυτό εν μέρει θα επιτευχθεί και μέσω των αναδιαρθρώσεων και μέσω της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής εξυγίανσης. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αν έχουμε ε, αυτή την μείωση στην αξιοπιστία και στην φερεγγιότητα σε ορισμένες από αυτές χώρες λόγω της ε, καθυστέρησης ε, στην εξυγίανση ή σε, με κάποιον τρόπο στη μείωση της φερεγγιότητας, αυτό θα επηρεάσει το κόστος δανεισμού. Επηρεάζει και τον δημόσιο προπολογισμό αλλά και τον ιδιωτικό τομέα μέσω της αύξησης του κόστους δανεισμού. Ευχαριστώ για τους ε, σοσιαλιστές, Λίεμ Χονγκόκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και στις 5 ε, Δεκεμβρίου σας απέστειλα δύο ε, γραπτές ερωτήσεις ε, για τον κανόνα 118 σε ό,τι αφορά τα ε, ωφέλη της ΕΚΤ που στη συνέχεια δόθηκαν στις εθνικές κεντρικές τράπεζες που το μετέδωσαν στις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό ε, συνάδει με το 123.1 της συνθήκης. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ποσό και την αξιοποίηση του χρόνου ε, ε, που δίνεται στις, στις τράπεζες για το ελληνικό χρέος. Δεν μου έχετε απαντήσει μέχρι τώρα, θα ήθελα παρακαλώ να απαντήσετε σήμερα. Ζητώ συγγνώμη αν ε, δεν λάβατε απάντηση. Μπορώ να σας απαντήσω σήμερα. Για το πρώτο. σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ομόλογα και τα, τα έσοδα που έχει η ΕΚΤΑ από αυτά τα ομόλογα ε, αποτελούν τμήμα του καθαρού ωφέλους της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας που διανέμεται σε όλες τις ε, ε τράπεζες, σε όλες τις τράπεζες βάσει τη, της κλίδας κατανομής. Οποιοδήποτε όφελος αυτό ε, γίνεται τμήμα του καθαρού ωφέλους της Εθνικής ε, Τράπεζας και αυτά διανέμονται στους ε, αντιστοίχους ε, μετόχους βάση των ισχυών κανόνων. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα δίνει στι εθνικέ κεντρικέ τράπεζε και εκείνοι, αν έχουν κάποιον νόμο ή άλλο εθνικό κανόνα, τα διανέμουν αυτά τα κέρδη στου δικού του μετόχου. Μπορεί να είναι κυβερνήσει ή όχι. Οι κυβερνήσεις λοιπόν ε, των κρατών μελών <laughs> είναι αυτές που αποφασίζουν πώς θα αξιοποιήσουν ε, τα κέρδη που λαμβάνουν από τις ε, επιμέρους κεντρικές τράπεζες συμπεριλαμβανομένες και οποιασδήποτε άλλη στήριξη και από άλλες και από άλλα κράτη-μέλη. Επομένω, οι, οι κυβερνήσει αποφασίζουν πώ αξιοποιούν αυτά τα κέρδη. Στην δήλωση της 27ης Νοεμβρίου 2011, το Eurogroup είπε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν να εξετάσουν μια δέσμευση για να περάσουν στον ε, συσσωρευμένο λογαριασμό της Ελλάδας ένα ποσό που θα ε, αθρίζεται στην Εθνική Κεντρική Τράπεζα ε, και θα στηρίζεται και στα συμπεφωνημένα μέτρα. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα στα αριθμητικά στοιχεία, όμως θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα της ΕΚΤ για το 2012 καθώς και ένα ε, τύπου θα δημοσιευθούν στις 21 Φεβρουαρίου 2013. Όλα αυτά λοιπόν θα ακουστούν δημόσια. Το δεύτερο, συγγνώμη, αλλά για το ποσό και την ε, χρησιμοποίηση της λανθάνουσας υπεραξίας ε, της ΕΚΤ καθώς ε, αγόρασε στην δευτερεύουσα αγορά, δευτερογενή αγορά και είχαμε περίπου 15 δις ευρώ εκεί πέρα. τι έγινε με όλα αυτά. Uh, um, I'm Απάντησα στο ερώτημα. Απάντησα και στις δύο ερωτήσεις. Συγγνώμη. Θα μοιραστεί σε όλες τις ε, εθνικές κεντρικές τράπεζες οι οποίες θα το μοιράσουν με βάση την εθνική τους νομοθεσία στους ε, μετόχους που μπορεί να είναι κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις θα αποφασίσουν στην συνεχεία αν θα δώσουν αυτά τα ποσά στην Ελλάδα ξανά ή όχι. Uh, Αν ζητάτε για την υπεραξία, ε, τα κέρδη για τα οποία μιλούσα ε, ε, συμπεριλαμβάνει και την υπεραξία αυτή. Έχω 45 δευτερόλεπτα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την λανθάνουσα υπεραξία, τη διαφορά ανάμεσα στην ονομαστική αξία των τίτλων που εισπράτεται στο τέλος, όταν φτάσουν στο τέλος της διάρκειάς τους, και την αγοραία τιμή στην οποία αγοράστηκαν αυτοί οι τίτλοι. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί δεν αναφέρεται στα αποτελέσματα. Γιατί εκεί μιλάμε, ε, χρησιμοποιούμε όχι την υπεραξία, αλλά την ονομαστική αξία. 1,4 δηλαδή δισεκατομμύρια ε, υπεραξίας για το 12. Και στο τέλος, δηλαδή όταν λήξουν αυτοί οι τίτλοι, το ποσό αυτό θα έχει φτάσει στα 15 δις. Ναι, και τα δύο τα συμπεριλαμβάνουμε. Ούτω ή άλλω αυτά θα τα δημοσιεύσουμε σε τρει μέρε. Λίαμ, συγγνώμη. Ε, Κάνει αυτήν την ερώτηση τρει μέρε νωρίτερα. Από το Ελκ. Ο κύριο Φέο. Φέιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντράγη, θα ήθελα να ξεκινήσω με το να σας συγχαρώ και να σας πω ότι συμφωνώ με πολλές από τις τοποθετήσεις που κάνατε εδώ και φυσικά για τη σπουδαιότητα της προσαρμογής των δημόσιων ε, λογαριασμών. Προέρχομαι από μια χώρα, την Πορτογαλία, που υπήρχε μεγαλύτερη χρέωση σε σχέση με τα ε, συνετά πλαίσια. Και συμφωνώ επίσης και με τις τοποθετήσεις που κάνατε για τις επιπτώσεις ε, βραχυπρόθεσμα για αυτά τα προγράμματα προσαρμογών, για την ανάγκη <clears throat> να αντιμετωπίσουμε τα πλήγματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά την φορολόγηση για παράδειγμα και ότι δεν υπάρχει η θεωρία του ένα μέτρο μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες. Θα ήθελα να θέσω τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, ποια είναι η αξιολόγησή σας για την δημιουργία και ε, κατάρτιση των προγραμμάτων προσαρμογών. Ιδιαίτερα για τις χώρες εκείνες που υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους, όπως π.χ. η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Δεύτερον, αυτή τη χρονική στιγμή υπάρχουν δυνατότητες να τροποποιηθούν αυτά τα προγράμματα και να δούμε αν είναι δυνατόν να λυθούν ε, τα μέτρα εκείνα που είναι αναγκαία πρόθεσμα για μια πολιτική φορολόγηση ε, που θα είναι λιγότερο επιβαρυντική για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρο ότι κατάλαβα απόλυτα τη δεύτερη ερώτησή σα, Μπορείτε να επαναλάβετε. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να γίνουν τροποποιήσεις στα προγράμματα προσαρμογών που θα επιτρέψουν αυτές οι τροποποιήσεις ε, να μην έχουμε αρνητικά ε, αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα ώστε για παράδειγμα να έχουν φορολογικές πολιτικές ε, τα διαφορετικά αυτά κράτη που θα είναι πιο, θα δημιουργούν κίνητρα για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το κύριο θέμα και σημείο εδώ είναι αν συγκρίνουμε τη σημερινή τρέχουσα κατάσταση με την κατάσταση πριν από ένα χρόνο πρέπει να πούμε ότι η πρόοδος που σημειώθηκε σε όλα τα μέτωπα και σημεία είναι πάρα πολύ αξιοπρόσεκτη. Είναι ιδιαίτερα σημαντική σε όλα τα πεδία και στην ε, φορολογική εξυγίαση και στις ε, διαθροτικέ ε, μεταρρυθμίσεις και στον τραπεζικό τομέα για να επιδιορθωθούν τα όσα έγιναν με λανθασμένο τρόπο. Φυσικά αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Συνολικά όμως όλες αυτές οι χώρες, οι χώρες που έχουν εγγραφή σε αυτά τα προγράμματα. Οι χώρες που πιέζονται βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι βρισκόντουσαν πριν από ένα χρόνο. Και το βλέπουμε αυτό και από διάφορους δείκτες δεν το βλέπουμε ακόμα στο, ε, στη συνιστόσα της απασχόλησης ακόμα, αλλά βλέπουμε καλύτερους τρέχου, τρέχοντες ε, λογαριασμούς και ε, ισολογισμούς, ιδιαίτερα σε σχέση με κάποιες διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με μια χώρα και μια άλλη χώρα, όμως υπάρχει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και το βλέπει αυτό κανείς σημα, ε, σφαιρικά, συνολικά και σε σχέση και με την φορολογική εξυγίαση, ο ρυθμός και η ταχύτητα διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά και πάλι εδώ πάντα πρέπει να βλέπει κανείς ε, τα πράγματα μέσα σε με συγκεκριμένο αναλογικό τρόπο. Και βλέποντας το τι συνέβαινε πριν από καιρό σε σχέση με την Ευρωζώνη, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Η κρίση, η αξιολόγηση είναι λοιπόν αξιολόγηση για μεγαλύτερη αναγνώριση των ε, όσων επετεύθησαν και την ανάγκη να συνεχίσουμε επί της πορείας αυτής, να συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι και να ιδιαίτερα όσον αφορά και χώρες που ε, χωλαίνουν όσον αφορά τις διαθροτικές αλλαγές ε, θα πρέπει να δράσουν ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί και τα αρνητικά φαινόμενα. Το δεύτερο, για τη δεύτερη παρατήρηση που θα μπορούσα να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να συνεχίσω απαριθμώντας πολλές από τις βελτιώσεις που σημειώθηκαν και βλέπουμε. Για να σας δώσω μια σφαιρική ιδέα. Πέρυσι, αυτή την εποχή του χρόνου πέρσι, 19 και πάνω από ε, τις 100 της έκδοσης ομολόγων ε, προερχόντουσαν από τις ε, χώρες αυτές. Τώρα πάνω από 60% έρχονται, προέρχονται από αυτές οι εκδόσεις από τις περιφερειακές χώρες. Και η βάση των επενδύσεων έχει επεκταθεί, έχει διευρυνθεί σημαντικά δεν βλέπουμε μόνο να αγοράζουν ομόλογα ε, κρατικού χρέους ε, οι ε, τράπεζες και επιχειρήσεις. Αγοράζουν αυτά τα ομόλογα διαφορετικοί, διάφοροι επενδυτές και εκτός της ζώνης ευρώ. Και βλέπουμε στους λογαριασμούς της Ευρωζώνης ότι βελτιώνεται η κατάσταση λόγω των ροών, κεφαλαιακών ροών που υφίστανται από τον υπόλοιπο κόσμο και τις περιφερειακές χώρες προς τη ζώνη ευρώ. Θα μπορούσα να ε, συνεχίσω να παριθμώ αυτά τα στοιχεία. Ε, ο ευμετάβλητος χαρακτήρας όμως έχει μειωθεί σε σχέση με την κατάσταση. Ε, volatility δηλαδή μειώθηκε. Και βλέπουμε ότι μια χώρα έχει πάντα τη δυνατότητα να ανασχεδιάσει, να ανακαταρτήσει το πρόγραμμά της μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνηθεί προηγούμενα βέβαια με, τις, με τους πιστωτές της. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Όμως τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες έχετε εσείς τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Οι αγορές θεωρούν υπάρχει μια καλμία, μια νηνεμία μετά από τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε επανέλθει στα ουσιώδη πάλι πορεία προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση δηλαδή. Σε αυτή την πορεία ε, προετοιμασίας για το, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου που κανονικά θα έπρεπε να εγγύψει του θέσματος, ήσασταν τμήμα ε, της ομάδας των τεσσάρων. Τελικά όμως άλλαξε η μερίσια διάταξη και παραπέμφθηκε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα των τεσσάρων τελικά αυτή ε, η ομάδα των τεσσάρων διαλύθηκε. Αν δούμε τα θέματα της νομισματικής ε, και οικονομικής εποπτείας, θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να γίνουν όλες αυτές οι συζητήσεις χωρίς εσάς ή θεωρείτε ότι εδώ που φτάσαμε για την ε, Τραπεζική Ένωση αρκεί η συνεισφορά σας για αυτή την πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Εγώ είχα καταλάβει ότι θέλατε αυτός ο μηχανισμός ε, ε, επίλυσης των κρίσεων να λειτουργήσει πιο γρήγορα. Πώς ε, οργανώνεται το χρονοδιάγραμμα, το γραμμά σας, και την μεταβλητή σας αυτή γεωγραφία προς αυτή την πορεία για μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Uh, first Οι συνθήκες είναι σαφώς καλύτερες. Και αυτό ισχύει, έγινε λόγω του OMT και λόγω όμως των ε, κυβερνητικών δράσεων. Εάν δεν δοθεί μια πραγματική πίεση προς την δημοσιονομική εξυγίανση και τις ε, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις από τις κυβερνήσεις, δεν θα γινόταν πραγματικό OMT. Εμείς δημιουργήσαμε πραγματική ε, νομισματική ένωση. Το 2013 θα είναι μια χρονιά εφαρμογής των αποφάσεων. Για διάφορους λόγους που τους ξέρετε καλύτερα από μένα. Η εφαρμογή είναι κλειδί. Πολλά πράγματα έχουν αποφασιστεί. Τώρα πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Η ΕΚΤ λειτουργεί ε, για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, Και μετά θα βοηθήσουμε και την Κομισιόν για να σχεδιάσει ε, και την ε, ενιαία αρχή εξυγίανσης. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα δώσει ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Λόγω του μεγέθους του και της ταχύτητας με την οποία λειτουργήσε, ε, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Λειτουργήσε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Για την ομάδα των τεσσάρων κάνατε την ερώτηση. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου θα έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Και εμείς θα συνεισφέρουμε. Ανάλογα με τις ανάγκες, ανάλογα με το τι θα μας ζητήσουν να κάνουμε. Αλλά η επίσημη διαμόρφωση πούμε, αυτής της ομάδας είναι κατά τη διαφορετική από ό,τι ήταν πέρυσι η επίσημη σύνθεση και η κατανομή των καθηκόντων. Από το ΕΛΚ, ο Μάριο, Μάουρο, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερα της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, της πίστοσης που δίνεται στην πραγματική οικονομία. Άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις που κάνατε για τις δυσκολίες που υπάρχουν για να περάσουμε από την τακτοποίηση ας πούμε των, του πλαισίου, ε, της χρηματοδότησης των τραπεζών ας πούμε και εν συνεχεία ε, η χρηματοδότηση από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Η ΕΚΤ πιστεύει ότι θα γίνει χρηματοδότηση προς τις τράπεζες ανάλογα με το αν έχουν προσανατολισμό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι αξιολόγηση κάνετε εσείς. Ε, τι μοντέλα δανεισμού έχουν όπως το funding for landing του, της, Ευρωπαϊκής, συγγνώμη, της ε, Βρετανικής Κεντρικής Τράπεζας. Um, the... Όπως Όπως, όπως προανέφερα, προβληματιζόμαστε διαρκώς ε, και συνεχώς γι' αυτό για αυτές τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την πολιτική μας. Πιστεύουμε ότι ήδη κάναμε πολλά. Υπό έναν όρο κάναμε κάτι ανάλογο όσον αφορά το funding for lending. Όταν είπαμε στις τράπεζες ε, μπορείτε τα δάνεια αυτά ως ε, ε, εγγύηση για περαιτέρω δανειακές και πιστοτικές πράξεις να τα θεωρήσετε. Σε σχέση λοιπόν με το κόστος ε, ή τη δράση της ε, Βρετανικής Τράπεζας, κάτι ανάλογο είναι. Τουλάχιστον θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Και όπως είπα προηγούμενα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για όρους και προϋποθέσεις. Αν εξαναγκάσουμε τράπεζες ε, να δανείζουν ε, τους ε, λανθασμένους ε, δανειοδότες τότε θα μπορεί να πάει κάτι στραβά αν δεν μπορούν οι δανειολήπτες να επιστρέψουν τα δάνειά τους, να αποσβέσουν τα δάνειά τους και οι τράπεζες πτωχεύσουν. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη ότι έχουμε 17 κράτη-μέλη στην Ευρωζώνη η εποπτεία αυτών των ε, προγραμμάτων όπου θα πρέπει να εποπτεύουμε και να ελέγχουμε ποια τράπεζα δανείζεται ώστε να διαθέσει πιστώσεις και δάνεια. Είναι πολύ πιο περίπλοκο το πλαίσιο δράσης από ότι μόνο σε μια χώρα συνολικά. Συγγνώμη τώρα που μίλησα αγγλικά. Okay, uh, did you wish Θέλετε να επανέλθετε εσείς με επερώτηση. No, okay. can uh, to... Τότε μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε στον κύριο Ντανίτσι ε, από πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από την Ιταλία. Όχι γιατί είμαι επαρχιώτης και κολλάω στην Ιταλία, αλλά γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ιταλία είναι στο κέντρο της προσοχής των Ευρωπαίων. Ειδικά μετά την ε, ε, θλιβερή αυτή η ιστορία της ε, τράπεζας της Σιένας. Νομίζω ότι το ε, Ιταλικό τραπεζικό σύστημα έλεγε τα ίδια και τα ίδια, κάποια πράγματα που το καθησύχαζαν το ίδιο, ε, θεωρούσε ότι είναι πολύ καλύτερο από άλλα τραπεζικά συστήματα, ότι είχε αντισταθεί πολύ καλύτερα από, άλλες, από άλλα τραπεζικά συστήματα, κάτι που δεν ίσχυε. Ενώ είδαμε ότι στην πραγματικότητα έχουμε και εμείς τέτοια προβλήματα. Τελικά τα ίδια συνέβησαν και στην Ιταλία. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα ε, ρύθμισης στην Ιταλία όσον αφορά ας πούμε, το ρόλο των Ιδρυμάτων και σε σχέση με το ρόλο των Ιδρυμάτων. Ποιος είναι ο ρόλος ε, του Υπουργείου Οικονομίας για αυτά. Τι γίνεται με τα περιουσιακά στοιχεία των Ιδρυμάτων. Εσείς μας μίλησατε σήμερα ε, για την ε, Τραπεζική Ένωση, μας μιλήσατε για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό κτλ. Πώς παντρεύονται αυτά τα δύο. Δεν θέλω να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσατε που είναι πολύ Ιταλο-Ιταλικά και δεν θέλω να μπω. Αλλά υπάρχουν δύο φάσεις. Το πώς ας το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα ανταποκρίθηκε στην κρίση. Το τραπεζικό σύστημα έδειξε σταθερότητα. Δεν χρειάστηκε να περάσει σε δημόσια ανακεφαλαιοποίηση. Αντίθετα από ό,τι συνέβη με πολλές άλλες χώρες και τις τράπεζές τους. Υπάρχει βέβαια ε, η μεμονωμένη περίπτωση αυτής της τράπεζας της Σιένας, της Μόντε Πάσκη, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα, εγκληματική δραστηριότητα κτλ. και ο ρόλος των τραπεζών κτλ. Εν συνεχεία, η αντίδραση του Ιταλικού τραπεζικού συστήματος αλλά και άλλων χωρών ε, στην παραδεταμένη κρίση είναι η επόμενη φάση. Και εκεί βλέπουμε ότι όταν έχουμε χαμηλά επιτόκια, από την άλλη όμως οι δυσχέρειες στην Ιταλία αυξάνουν, τότε δείχνει τις δρογμές στο Ιταλικό σύστημα. Ε, οι μεγάλες τράπεζες βέβαια έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση. Η Monte di χρειάστηκε μία έχηση κεφαλαίου γιατί το χαρτοφυλάκιο των τίτλων ε, ε αξιοποιείται με βάση τον, ε, τις τιμές που είχε τον Ιούνιο του 2011. Γενικότερα το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα δείχνει όπως και άλλα συστήματα, την έκθεσή του στην παρατεταμένη ε, ύφεση. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει. Εν πάση περιπτώσει, τούτου λεχθέντος, οι μεγαλύτερες τράπεζες έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση. Παρότι εδώ και δύο χρόνια, ενάμιση τέλος πάντων χρόνο έχω φύγει από την ε, Ιταλία και δεν ξέρω τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, η κεντρική Ιταλική τράπεζα είναι αυτή η οποία έχει το, το βασικό ρόλο εδώ να παίξει. Τον ηγετικό ρόλο. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Εγώ ήθελα να σας πω ότι πρόσφατα ε, είπα όλα αυτά τα θέματα, αναφέρθηκα σε όλα αυτά τα θέματα που αναφερθήκανε και από τον α, διοικητή της Ιταλικής Τράπεζας. Κοιτάξτε, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά δεν θέλω να ασχολιάσω καθόλου το θέμα των ιδρυμάτων στην Ιταλία. Ευχαριστώ. Ελκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα Σουηδικά, σε ελεύθερη μετάφραση, έχουμε μια παροιμία. Μην πείτε, ε, μην, μην λέτε αντίο μέχρι να έχετε περάσει το ουράνιο τόξο. Και αυτό είναι σημαντικό εδώ πέρα, σε αυτά τα στοιχεία τη ανάκαμψη. Ε, αναφερθήκατε σημαντικά στοιχεία, όπω είναι το εργατικό κόστο, άλλε αλλαγέ ε, σε ό,τι αφορά του εμπορικού λογαριασμού και το καθεξή. Όμω, μεγάλο αριθμό μεγάλων οικονομιών βρίσκονται σε ένα είδο ε, ύφεση και με δυσμένες προοπτικές. Υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική πολιτική και πώς ε, κάποια κρατημέλη θα μπορέσουν να υλοποιήσουν ε, το νέο πακέτο σταθερότητας ε, και δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντοπίζετε εσείς ό,τι αφορά τη δημοσιονομική σταθερότητα για κάποιες ελλείψεις, αδυναμίες και πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε. Αυτή είναι η ερώτηση με το μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Αυτό που είπα είναι ότι υπάρχουν ενδείξεις βελτιωμένης δημοσιονομικής σταθερότητας στον χώρο του ευρώ και ανάκτησης της εμπιστοσύνης. Και αναφέρθηκα σε μια σειρά παραγόντων που θα δώσουν πραγματική ουσία σε αυτή τη δήλωση. Όμως, πράγματι υπάρχει ε, μια αδυναμία. Και η κατάσταση θα παραμένει ευάλωτη έως ότου δούμε σταθερότητα. Πρέπει να δούμε, ε, ανάπτυξη, συγγνώμη, πρέπει να δούμε ε, αύξηση των κεφαλαϊκών ροών. οι κίνδυνοι για την οικονομική δραστηριότητα βρίσκονται ακόμα σε δυσμενή επίπεδα λόγω της υψηλής ανεργίας, της χαμηλής κατανάλωσης και των χαμηλών επενδύσεων. Επομένως δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Το έχω πει στο παρελθόν και δεν έχω λόγο να αλλάξω αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στην ε, διόρθωση ε, των συλλογικών μας συλλογισμών και των ε, κρατικών και των τραπεζικών και να επιδιορθώσουμε τις κεφαλαιογορές μας στην χώρο, στο χώρο του ευρώ. Πολλά από τα ζητήματα που μου έχετε θέσει αφορούν ακριβώς αυτό, την επιμονή και την διατήρηση του κατακαιρματισμού. Κάποιο είπε γιατί πρέπει οι ίδιε μικρομεσαίε επιχειρήσει να πληρώνουν ε, διαφορετικά επιτόκια. Αυτό είναι ένα από τα βασικά εμπόδια ε, στην ε, ανάκαμψη και στην ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά παραπάνω αυτή τη στιγμή. Επομένω, οι δυσκολίε παραμένουν, πρέπει να συνεχίσουμε και να επιμείνουμε και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την αλλαγή της διακυβέρνησης ε, της Νομισματικής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. I think this was very... Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας συνιστούσα να θυμόσαστε αυτό το απόφθεγμα, το σουηδικό απόφθεγμα βλέποντας ε, τα τελευταία χρόνια υπερβολικά πολλές φορές είπαμε τα καταφέραμε και δεν τα είχαμε καταφέρει, δεν είχαμε ξεπεράσει τα προβλήματα και υπάρχει βέβαια ανάγκη να είναι κανείς αισιόδοξο και να αξιολογεί θετικά τα κεκτημένα και αυτά που έχει επιτύχει αλλά και ρεαλιστικά να μπορεί να σκέπτεται για την ανάγκη να υπάρχουν και άλλες ε, μεταρρυθμίσεις ε, και άλλες αλλαγές που πρέπει να ακολουθήσουν. Καμιά φορά είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι ε, αξιολογώντας τα προβλήματά μας και σε αυτή τη χρονική στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε με αυτόν τον τρόπο να εστιαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ρεαλιστική αξιολόγηση της κατάστασης όσοι υφίσταται και χρηματοοικονομικά και από πλευρά των τραπεζών και της, των ίδιων των αναγκών που υφίστανται προτού πούμε τα καταφέραμε. Και τώρα για από πλευρά της Άλντε Όλε Σμιτ παρακαλώ. Συγγνώμη πρόεδρε. Είναι κάπως πιο εθνικιστική εστίαση από πλευρά των Σκανδιναβών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί η Δανία και η Σουηδία θα έπρεπε να ενταθούν στο ευρώ. Διαβάσατε φυσικά σε σχέση με το άρθρο αυτό στο περιοδικό Economist. Και λένε και ε, κάποιοι σε σχέση με την ε, ε, ανάγκη να ενταχθούμε στο ευρώ, αλλά βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα. Το ευρώ είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Και τα διαφορετικά νομίσματα λένε άλλοι ότι είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν αληθεύει αυτό. Ίσως όμως κάποιοι δεν με ακούν. Εσείς ίσως θα μπορούσατε να δώσετε κάποια σχόλια για να πιστούν. Είναι θεμελιώδους σημασία αυτά. Διότι Άλλε χώρε θέλουν να ενταχθούν στη ζώνη ευρώ και δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει την κρίση. Και για τι ε, νέε προτάσει ε, που υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρηματοοικονομικό πλαίσιο δείχνουν ότι είναι ένα πρόβλημα να είναι κανείς εκτός της Ευρωζώνης. Πιστεύετε ότι αυτή η αρχή της ε, ε, δυνατότητας ε, έκδοσης ή του να είναι κανείς μέλος είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και πώς θα μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα όταν εταιρείε εκτός Ευρωζώνης αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω του ότι είναι εξοεδαφική η εφαρμογή αυτών των αρχών για αυτές και αυτό είναι ένα ειδικό πρόβλημα για χώρες αντιδική μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το πρώτο σας ερώτημα. Είμαι προκατηλημένος. Θεωρώ ότι το ευρώ είναι κάτι το πολύ θετικό και καλό. Και οπωσδήποτε θα πρέπει από κοινού να μπορέσουμε να, ε, να έχουμε μια δυνατότητα ευημερίας. Διότι διαφορετικά θα είμαστε όλοι θύματα αυτής της κρίσης αν δεν ε, κάνουμε αυτά τα οποία είναι αναγκαία. Για παράδειγμα, πόσα διάφορες χώρες με διαφορετικά νομίσματα και διαφορετικές ε, ισοτιμίες θα είχαν αντιμετωπίσει την ε, χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Η απάντηση που δίνεται είναι ότι η αστάθεια που θα απέρεε θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από την κατάσταση που είχαμε στην Ευρωζώνη με το ενιαίο νόμισμα, με το ευρώ. Είμαι βέβαια προκατηλημένο υπέρ του ευρώ, αλλά η απόφαση τελικά να ενταχθεί κανεί στη ζώνη ευρώ βρίσκεται στα χέρια απόλυτα των ε, αρμόδιων κυβερνήσεων που κυρίαρχα αποφασίζουν από πλευράς τους. Ε, δεν θέλω να πείσω κάποιες χώρε που βρίσκονται εκτός ευρώ να ενταχθούν στη ζώνη ευρώ οπωσδήποτε. Δική τους υπόθεση είναι, αλλά ε, υπάρχουν πολλά ωφέλη από το ευρώ και μπορούν να αποκομίσουν πολλά ωφέλη από το να ενταχθούν στο ευρώ. Για παράδειγμα σε σχέση με, το, με τις διαστάσεις της, ε, ε, των ΙΠΑ έχουμε σταθερότητα νομισματική που δεν είχαμε στο παρελθόν για πολλές χώρες. Μην το ξεχνάμε. Έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια ιστορικά αυτή τη χρονική στιγμή. Πολύ εύκολα ξεχνά κανείς αυτή τη στιγμή τον μεγάλο κατάλογο των ε, θετικών κεκτημένων και ωφελημάτων ε, που απέρευσαν από τη ζώνη ευρώ. Τώρα, σε αυτή τη χρονική συγκυρία με την ε, οικονομική κρίση και τον υπερβολικό βαθμό ανεργίας των νέων, βλέπουμε όμως ότι έχουμε και από την άλλη πλευρά και κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν θα είχα όμως τις ε, γνώσεις για να σχολιάσω όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε. Με κάθε σεβασμό συνεχίζει ο κύριος Σμιτ γιατί πρόκειται για την Ευρωβουλή για ένα ε, κατεξοχήν πολιτικό σώμα και γι' αυτό διατυπώνουμε και πολιτικά ερωτήματα. Είναι κέρια σημασία να ακούμε τις απόψει σας, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εσείς είσαστε οι πιο αξιόπιστοι και εσείς ο πιο αξιόπιστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ή άλλω. Η αλλω η ερωτηση μου αφορά αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι δεν θα έπρεπε λέτε να πείσετε. Το αντίθετο, άτομα όπως εσείς θα πρέπει διαζώσεις να αναφέρετε τα επιχειρήματα για να μπορέσετε να πείσετε κάποιους. Αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερο στη σημερινή συγκυρία. Πρέπει να ακούσουμε τα θετικά επιχειρήματα. Γιατί πρέπει να, να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να παγιωθεί η ζώνη ευρώ. Διότι θα είναι το κοινό μας πεπρωμένο, η κοινή μας πορεία και πρέπει και οι Σκανδιναβοί να τα ακούσουν και να τα λάβουν υπόψη από πλευρά σας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυτά. Θα το πάρω αυτό το οποίο εσείς μου δώσατε ως μήνυμα, αυτό αποκομίζω από αυτή τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στο ΕΛΚ. Γκέι Μίτσερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη. Η Ιρλανδία δεσμεύτηκε να ε, εξασφαλίσει βιώσιμα δημοσιονομικά. Από το 2008 έχουμε ολοκληρώσει την δημοσιονομική εξυγίανση αξίας 30 δισεκατομμύρων ευρώ που είναι το 30% του ΑΕΠ μας. Ε, οι διευθετήσεις που έγιναν για την ανταλλαγή των γραμματείων έχει πέσει τώρα η αξία τους. Οι αναλυτές είπαν ότι το Ιρλανδικό Δημοσιονομικό Σύστημα και όλη η Ευρωζώνη θα υποφεληθεί με μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια λόγω της ε, διευθέτησης και μείωση ε, και θα μειωθεί ε, η χρηματοδότηση που χρειάζεται η Ιρλανδία. Η ΕΚΤ θα κοιτάξει, θα ξαναεξετάσει αυτή τη διευθέτηση και η ΕΚΤ θα εξετάσει όλα όσα, τα, όλα όσα μέτρα χρειάζονται, ώστε να λειτουργήσουν καλά τα πράγματα και όλα όσα εμπίπτουν στην εντολή της. το ερώτημα στα σχόλιά σας στις 7 Φεβρουαρίου, την μέρα που ανακοινώθηκε αυτή η διευθέτηση, αναφερθήκατε σε αυτή τη διευθέτηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ιρλανδικής ε, Κυβέρνησης και είπατε ότι το Δουσού ομόφωνα σημείωσε α, το πώς έχει αυτή η συμφωνία. Θέλω να ενημερώσετε την Επιτροπή αν υπήρξε καμία ουσιαστική αλλαγή σε αυτή τη θέση από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και θεωρώ ότι δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή θέσης. Well, Σωστό είναι αυτό, κύριε Μόντι. Τι σημαίνει έγινε ή δεν έγινε αλλαγή. σε κάτι που απλώς σημειώνουμε ότι συνέβη. Μάθαμε, ενημερωθήκαμε για, την, για το ότι έλαβε χώρα. Δεν μπορούμε μία εβδομάδα μετά να πούμε «Α, δεν ενημερωθήκαμε». Όχι. Το σημειώσαμε. α πώς μπορώ να αλλάξω τη θέση μου, η οποία θέση είναι... Ε, το σημειώνω. Δεν είπα ότι το εγκρίνω ή δεν το εγκρίνω. Επομένως, ε, επιμένετε στο σημείωμα που αρχικά είχατε... Ε, ή μάλλον, ε, επιμένετε στην αρχική σας δήλωση, που, που, η οποία ήταν πια, το σημειώνουμε. Σημειώνουμε αυτή την ε, συμφωνία μεταξύ της α, ε, κυβέρνησης και της α, ε, Κεντρικής Τράπεζας. Ποια είναι η προοπτική του ευρώ, κύριε Ντράγκη, και με βάση την, την, τις επιδόσεις της Ιρλανδικής οικονομίας πιστεύετε ότι η Ιρλανδία θα απαλλαγήσει ως νούπο από το πρόγραμμα με βάση τις επιδόσεις που είχαμε, τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Πιστεύετε ότι είναι πιθανό σύντομα να βγούμε από το πρόγραμμα, να μην έχουμε πλέον ανάγκη το πρόγραμμα ως χώρα. Δεν μπορώ να το προδικάσω. Αλλά η Ιρλανδία ακολούθησε την προδιαγεγραμμένη πορεία ε, ως προς το πρόγραμμα. Σε όλα, ως προς τα, όλα τα τμήματα του προγράμματος, με μεγάλη επιτυχία και οι επιδόσεις ε, ήταν πολύ σημαντικές. Υπάρχουν τμήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα που χρειάζεται περαιτέρω δράση, σίγουρα. Αλλά γενικά είναι μια χώρα η οποία τα πήγε αξιοθαύμαστα. Πιστεύω λοιπόν ότι το πρόγραμμα ε, εκπνέει στο τέλος του 2013 αν δεν απατώμε, και εν συνεχεία θα κάνουμε μια αποτίμηση. Αν μπορώ να μιλήσω κι εγώ για την Ιρλανδική κατάσταση. Είναι σωστό. Σημειώσατε. Ε, Επομένως δεν έχετε την να, να φέρετε αντίρρηση τώρα θα εκδοθούν δηλαδή τα ομόλογα και θα επιστρέψουν στις αγορές τα ομόλογα αυτά. Αυτό σημαίνει το γεγονός ότι εσείς σημειώσατε τη συμφωνία. Με βάση το άρθρο 113 θα αξιολογήσουμε τη συμμόρφωση, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Και εκείνη την ε, χρονική στιγμή θα δούμε εάν η συμφωνία, τέλος πάντων, η συναλλαγή μεταξύ της ε, Ευρωπαϊκής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 113. Και αν όχι θα δούμε τι άμεση νομική δράση πρέπει να λάβουμε. Ευχαριστώ ε, για αυτή τη διευκρίνηση. Ο Πίτερ ε, Σάιμον. Μάλιστα κύριε Ντράγκη, ερώτησή μου, ερώτησή μου που στοχεύει Πώς εμείς στην ανταλλαγή αυτή των απόψεων μαζί σας θα μπορούμε να φανταστούμε όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο τέλος τέλος θα είναι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Ήδη σήμερα έχουμε αυτή την κατάσταση ότι ο κανονικός απλός πολίτης, ε, φυσικά νομικά πρόσωπα για την πρόσβαση στα έγγραφα της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν πρόσβαση υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται, ε, δεν υπονομεύεται το κοινό συμφέρον. Υπάρχει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρόσφατα ότι δύο μελέτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα δεν μπόρεσαν να δημοσιοποιηθούν ε, με, την αιτιολόγηση ότι Προ προστασία του κοινού συμφέροντος όσον αφορά την νομισματική και οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας που θα υπονομευόντουσαν αν δημοσιευόντουσαν. Λοιπόν, εδώ δημόσια ανταλλάσσουμε απόψει όταν θα έχετε τον εποπτικό αυτό ρόλο και ιδιαίτερα όσον αφορά τα συστημικά ε, ε, σημαντικά όργανα όταν θα πρόκειται για την άσκηση των ε, δικών σας, κυριαρχικών δικαιωμάτων, εποπτικών δικαιωμάτων, όταν κάτι το συστημικό θα διαπιστώνεται. Πάλι σε τακτή βάση το κοινό συμφέρον θα βρίσκεται στο πεδίο έντασης ε, στο, σε σχέση με το δικό μας δικαίωμα να ενημερωνόμαστε και να είναι όλα αυτά δημόσια. Πώς βλέπετε την ανταλλαγή απόψεων και, και πρόσβαση σε τέτοιου είδους έγγραφα τον δικό σας ρόλο όταν θα είσαστε η εποπτική αρχή. Πού βρίσκεται το όριο για την λογοδότηση από πλευρά σας ε, και σε σχέση με την προστασία του κοινού συμφέροντος όταν θα συναλλάσσεστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντράγκη. Υπάρχουν δύο διαφορετικές πτυχές στην ερώτηση. Η πρώτη είναι η λογοδοσία. Και αυτό πραγματικά αφορά τον νομοθέτη και το κοινοβούλιο. Το μόνο που μπορώ να πω επ' αυτού είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πρόθυμη να λογοδοτεί σε όλα τα πλαίσια και με κάθε τρόπο. Και οπωσδήποτε ο επιμερισμός ε, των αρμοδιοτήτων, εποπτικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την ανάγκη λογοδοσίας από πλευράς μας έναντι των άλλων. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα υπήρχε καμία αντίρρηση στο να υπάρξει αυξημένη λογοδοσία. Θα είμαστε απόλυτα πρόθυμοι και να δεσμευτούμε να το διασφαλίσουμε αυτό. Τώρα, να το, να το αποφασίσουμε αυτό πότε και πόσα θα βρίσκεται και στη διακριτική ευχαίρεια και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Τώρα, για τα θέματα διαφάνειας. Αναφερθήκατε στην ε, ε, περίπτωση Bloomberg και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ σε σχέση με διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρέπει να διατηρήσουμε, να διασφαλίσουμε την εξή πτυχή. Η νομισματική πολιτική και η εποπτεία πρέπει να διαχωρίζονται αυστηρά μεταξύ τους. Και για τους λόγους, ε, για τη στάση που τήρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως νομισματικό όργανο, σε σχέση με τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση που αναφέρθηκε, μπορεί αυτό να μην συμβαίνει και να μην ισχύει όταν θα έχουμε τον εποπτικό ρόλο, όταν θα είμαστε το Ευρωπαϊκό Εποπτικό Όργανο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί όμως για το SSM να ισχύουν και όχι για την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπό το νομισματικό πρίσμα. Πρέπει με αυτές τις διαχωριστικές γραμμές να εστιαστούμε σε αυτό και να μπορέσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα όταν θα έρθει η ώρα να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. we can press Προχωρούμε. Τελευταία ερώτηση, και από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ για τα όσα είπατε για το άνοιγμα του μηχανισμού ε, της του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Αν πρέπει να αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή Τα κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης θα πρέπει να προσδιοριστούν ως μέλη της Ευρωζώνης με προσωρινή απαλλαγή. Εφόσον υπάρχει αυτή η δέσμευση της συνθήκης, συνδέονται τα νομίσματά τους με το ευρώ και είναι απλώς θέμα χρόνου η προσχώρησή τους. Δεν είναι λοιπόν λογικό να βγάζουμε αυτές τις χώρες εκτός του νέου οικοδομήματος. Από αυτή την πλευρά λοιπόν θεωρώ ότι στα βάθη της καρδιάς σας κύριε Ντράγκη είστε τραπεζίτης όλων των Ευρωπαίων και όχι μόνο των μελών της Ευρωζώνης. Ε, στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού έχουμε το πρόβλημα της ε, εποπτείας ε, για τα κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης. Βρέθηκε μια μη τέλεια λύση αν θέλετε, αλλά εάν αυτά τα μέλη, αυτά τα κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης ε, δεν επιτραπεί να συμμετέχουν στον ESM, τότε θα υπάρχει εποπτεία χωρίς ε, μηχανισμό ε, διάσωσης, χωρίς αυτό το δίχτυ ασφαλείας. Έτσι θα δημιουργηθούν δύο κατηγορίες τραπεζών υπό τον εποπτικό μηχανισμό. Αυτές που θα τη χάνουν εποπτείας, αλλά και θα λαμβάνουν στήριξη η διάσωση και οι άλλε που απλώς θα τη χάνουν εποπτείας, θα τους λέει ο εποπτικό μηχανισμός τι να κάνουν και θα, θα τους αφήνουν στην τύχη τους. Έτσι έχουμε ανισότητες μέσα σε έναν νέο τραπεζικό χώρο. Να σας υπενθυμίσω ότι σε αυτές τις χώρες εκτός ευρωζώνη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ε, πάνω από το 70% των τραπεζών ε, ε είναι σε ιδιοκτησιακό καθεστώς μητρικής τράπεζας. Σήμερα τι βλέπουμε, ότι δεν έχουμε κρίση του ευρώ ως νομίσματος, αλλά της υπερχρέωσης κρατών και τραπεζών. Κάποιες από αυτές είναι στην Ευρωζώνη, κάποιες εκτός. Και αυτό το ξεχνάμε κάποιες φορές. Έτσι, είναι λάθος και παράλογο να περιορίζουμε ε, αυτό το οικοδόμημα και τα μέτρα που λαμβάνουμε μόνο στην Ευρωζώνη. Γιατί να το κάνουμε, είναι πιο εύκολο, είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο επίπεδα αλληλεγγύης ε, μέσα στην Ένωση. Και πέραν αυτού, ε, στο βιβλίο της Σελβί Γκουλάγ που παρουσιάστηκε προσφάτως και του Μάριου Μόντι, γίνεται λόγος για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Ευρωζώνης, που βεβαίως και σοκάρει οποιονδήποτε είναι εκτός Ευρωζώνης. Ε, δημιουργεί σοβαρές οικονομικές εστρεβλώσεις, παραβιάζει ε, κανόνες ανταγωνισμού ε, στην Ευρώπη και τα μέλη εκτός Ευρωζώνης, αν δεν τους επιτραπεί να συμμετάσχουν ισότιμα σε αυτό τον μηχανισμό και αν πληγούν, θα πρέπει να αναλάβουν μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν την ολοκλήρωση ε, της ενιαίας αγοράς. Έτσι πρέπει να βρούμε ανοιχτές ε, λύσεις χωρίς αποκλεισμούς ε, στις μελλοντικές μας προσπάθειες. Τα επόμενα βήματα το, ο ενιαίος ε, μηχανισμός εξυγίανσης, το σύστημα ε, διασφάλισης των καταθέσεων και πού αυτά τα κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης θα βρουν τη θέση τους στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού. Ευχαριστώ. Κύριο Στράγκη, το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι η κατεύθυνση που έχουμε ακολουθήσει όλοι μαζί λογικά κατά τη δημιουργία του SSM. Ξεκινήσαμε με την δημιουργία των θεμελίων αυτής της Τραπεζικής Ένωσης. Ο πρώτος στόχος που θέλουμε να επιτύχουμε είναι ουσιαστικά να επανέλθουμε στην κατάσταση μετά την κρίση. Τι είδαμε εκεί, ότι αν όχι πολύ, αρκετοί μεγάλοι, με, μεγάλοι ε, διασυνοριακοί θεσμικοί φορείς ε, πτώχευαν. Από εκεί λοιπόν φάνηκε η ανάγκη για μια πολύ πιο ενισχυμένη συνεργασία, συντονισμό και εποπτεία. Συλλογικά λοιπόν καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στον χώρο της Ευρωζώνης προκειμένου να έχουμε μια ε, νομισματική ένωση με μεγάλες συστημικές διασυνοριακές τράπεζες, για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε ε, μία ενιαία εποπτική αρχή. Στη συνέχεια ανακαλύψαμε ότι από την κρίση φαινόταν και κάτι άλλο. Ότι υπήρχε ένας στρεβλός ε, συνδεσμός μεταξύ των ομολόγων και των τραπεζών. Και για να κοπεί αυτός ο δεσμός πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ε, μία ενιαία εποπτική αρχή της Ευρωζώνης. Για πολλούς ε, λόγους αυτή ήταν η συλλογική εκτίμηση ότι θα, το εποπτικό πλαίσιο θα είναι πολύ πιο δυνατό και εύρωστο αν υπάρχει ενιαία εποπτική αρχή. Βεβαίω και σε στενή συνεργασία με τι εθνικέ εποπτικέ αρχέ. Όμω η κύρια ευθύνη θα βρίσκεται στην κεντρική αρχή. Το τρίτο σημείο και βεβαίως ε, σκιαγραφίσαμε και τους υπόλοιπους ε, πυλώνες, ε, την ενιαία αρχή εξυγίανση, τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανση και το καθεστώς διασφάλισης καταθέσεων. Όμως, η εγγύηση καταθέσεων. Όμω από εκεί και πέρα κανένα δεν θέλει να καταστρέψει βεβαίω την ενιαία αγορά. Όλοι συμφωνούμε ότι η ενιαία αγορά είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μα. Και δεν αμφισβητούμε αυτό το επίτευγμα. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε να βρούμε λύσεις για αυτή την αντικειμενικά περίπλοκη κατάσταση. Γιατί 17 χώρες μοιράζονται ένα νόμισμα. Έχουν ειδικέ ε, ανάγκες ε, και με έναν ε, δικό τους ρυθμό. Όμως ο τελικός στόχος είναι η διατήρηση της ενιαία αγοράς. Πρέπει να πετύχουμε λοιπόν αυτά που θέλουμε για το ευρώ, ταυτόχρονα όμως να διατηρήσουμε την ενιαία αγορά. Κάνω κάτι λάθο, ε, Πρόεδρε, βλέπω ότι σημειώνεται. Είναι ότι έχουμε περάσει το χρονοδιάγραμμα για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Αλλά συνεχίστε. Όχι, ολοκλήρωσα την απάντησή μου. Σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμού μας ε, έχουμε πέντε λεπτά για την απάντηση ερωτήσεων το πολύ. Ναι. Αν επιτρέπετε, Σάρων, μια και αναφέρθηκα και δεν ήμουν η μόνη που αναφέρθηκε κάτι που είπε και όχι με το σωστό τρόπο. Θα ήθελα να πω αυτό το οποίο αναφέρω σε σχέση με αυτά τα οποία ε, αναφέρθηκαν στο βιβλίο είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε στην αρχή για την ένταξη στο ευρώ σε σχέση με την κατάσταση για εκείνους που βρίσκονται εκτός ευρώ και εκείνων που βρίσκονται εντός ευρώ. Δηλαδή να υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με αυτούς που έκαναν αυτή την επιλογή να βρίσκονται εκτός τελεσίδικα. Σε σχέση με τις ε, δυνατότητες ε, επιλογής ε, όσον αφορά τις διαβουλεύσεις για το SSM. Αυτό ολοκληρώνει το νομισματικό διάλογο για αυτά τα θέματα και συνεχίζουμε με την ακρόαση με τον ε, Μάριο ως ε, επικεφαλής ε, για τους συστημικούς κινδύνους ως αρμόδιο. Πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Προτείνω... Διάλειμμα πέντε λεφτά. Εσείς θα απεμπολούσατε την τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση λοιπόν διαγράφεται από πλευρά του ΕΚ. Θα έχουμε ένα ε, τεχνικό διάλειμμα πέντε λεπτών λοιπόν. 5 λεπτών διάλειμμα ε, που ζήτησε το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. I just want to say, read the book. Don't listen to people who have read the book in the past. We have read the books. Oh, all the books. I have. Right, well we have to start again because... Um... Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί ο πρόεδρος θα πρέπει να φύγει εγκαίρως για να προλάβει την πτήση του. Δεν ξέρω πού πηγαίνει, ίσως στη Φραγκφούρτη. Έχουμε τώρα τη δεύτερη εισαγωγή του Πρόεδρου Ντάγκη σε σχέση με το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων. Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά εμφανίζομαι στην Επιτροπή σας να σας ενημερώσω για τις δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Όπω ξέρετε, το καθήκον του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου είναι να εντοπίσει και να παρακολουθήσει το συστημικό κίνδυνο και να εκδώσει συστάσεις πολιτικής για το μετριασμό αυτών των κινδύνων. Σήμερα, με μεγάλη χαρά, θα παρουσιάσω δύο νέες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ESRB. Ένα για τον τρόπο μετριασμού κάποιων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στις δραστηριότητες χρηματοδότησής τους και ακόμα μία σύσταση για την ενίσχυση του ρυθμιστικού, κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την, τις χρηματαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για την τρέχουσα κατάσταση. Εν συνεχεία θα σχολιάσω τις νέες συστάσεις. Και στο τέλος θα ολοκληρώσω παρουσιάζοντας κάποιες προσπάθειες, κάποια δουλειά που κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη διασύνδεση και για το υγιές μακροπροληπτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω με κάτι θετικό σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των συνθήκων των χρηματαγορών του πρόσφατου μήνε. Τα spread των κρατικών ε, ε, ομολόγων απέναντι στη Γερμανία μειώνονται και ορισμένε χώρε όπω η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχουν εκδώσει μεσοπρόθεσμα κρατικά ομόλογα για πρώτη φορά από το 2010 και οι γενικοί δείκτες ε, του συστημικού κινδύνου υποχώρησαν σημαντικά. Επιπλέον, η γεωγραφική, ο γεωγραφικός κατακαιρματισμός τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβησης που έχει χαρακτηρίσει σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή κρίση χρέους ε, μειώνεται και οι ροές καταθέσεων αρχίζουν να σταθεροποιούνται καθώς και οι ανισορροπίες του στόχου 2 υποχωρούν σε σχέση με τα ανώτατα όρια που είχαν φτάσει στα μέσα του 2012 όπου ήταν Κοιτάξτε, ήμασταν φέτος σε περίπου 20% κάτω από τον Ιούλιο του 2011. Ε, Επιπλέον, οι αγορές ε, χρηματοδότης από τις τράπεζες έχουν δείξει σημάδια βελτίωσης, καθώς δείχνουν, ε, δείχνει και η διάθεση των επενδυτών για το τραπεζικό χρέος ευρωζώνης. Όμως, μια αδύναμ, κάποιες αδύναμες μακροοικονομικές προοπτικές για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να επηρεάσουν την κερδοφορία των τραπεζών και τα επίπεδα των κεφαλαίων. Ε, μπορεί οι τράπεζες να καταθέσουν τις, την απαραίτητη, να καθυστερήσουν συγγνώμη, την απαραίτητη απομόχλευση και την εκαθάριση των ισολογισμών τους και αυτό μπορεί να ε, δημιουργήσει πρόβλημα στις μακροοικονομικές σχέσεις και να δημιουργήσει δυσκολίες στο να βρεθεί κεφάλαιο και πίστοση ε, που θα πάει στην πραγματική οικονομία. Φυσικά ε, η αναζήτηση της απόδοσης ε, είναι αυτή που επιδιώκουν οι επενδυτές. Ε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που τους οθούν στο να παραμένουν ακόμα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε, υπάρχουν κίνδυνοι τους τελευταίους μήνες που έχουν ανακύψει και οι ευρωπαϊκές τράπεζες ε, έχουν ε, υψηλές ανάγκες ε, αναχρηματοδότησης και θα έχουν τα, επόμενα χρόνια και θα εξακολουθούν να, είναι, να εξαρτώνται πολύ από την κεντρική τραπεζική χρηματοδότηση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις από μακροπροληπτική προοπτική. Αυτό σημαίνει υποστήριξη μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη και βοηθούν την υγιή μακροοικονομική δυναμική Δεύτερον, να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να εκαθαρίσουμε τους ισολογισμούς των τραπεζών με βάση ένα διαφανή τρόπο, να εφαρμόσουμε επίσης μια προληπτική αποτίμηση των ε, ε, στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών και ένα ενισχυμένο συντονισμό για την αναθεώρηση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Τρίτον, να παρακολουθήσουμε του σύνεγγυ την πιθανή συσσόρευση ρογμών στι χρηματαγορέ, ούτω ώστε να ενισχύσουμε την αντοχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περίπτωση μιας κρίσης ε, και εδώ να λάβουμε υπόψη μα και ενδεχόμενους μηχανισμούς απορρόφησης κραδασμών και τέταρτον να ενισχύσουμε την παρακολούθηση των κινδύνων ε, για τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Για να σταθώ στο τελευταίο αυτό σημείο, θα ήθελα τώρα να, ακριβώς γι' αυτό να σταθώ στις δύο συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ε, δημοσιεύθηκαν σήμερα. Το ένα από, μια από αυτές αφορά την ενίσχυση ακριβώς της χρηματοδότησης των τραπεζών, την ενισχυμένη χρηματοδότηση της, ε, των τραπεζών. Να δούμε λοιπόν την πρώτη. Στη τελευταία κρόαση στην Επιτροπή σας είχα αναγγείλει ότι όταν επιστρέψω θα παρουσιάσω τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις, τα ευαίσθητα σημεία που συνδέονται με την χρηματοδότηση των τραπεζών και των περιουσιακών του στοιχείων. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν ακριβώς αυτή την σύσταση με βάση αυτές τις αξιολογήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στους κινδύνους που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και στις απαντήσεις που θα, θέλα, θέλαμε να δώσουμε. Καταρχάς, η δομή χρηματοδότηση παρουσιάσει ρογμέ ε, για πολλά από τα πιστοτικά μα ιδρύματα. Η κρίση έδειξε ότι βασίζονται πάρα πολύ σε ασταθή, ε, κεφάλαια και σε μια αλλαγή της διάρκειας ε, των τίτλων ε, πολύ έντονη. Για, ακριβώς αυτό το, για αυτό το λόγο ακριβώς οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου συστήνει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να υποβάλουν τα δικά τους σχέδια χρηματοδότησης στους εθνικούς, ε, στις εθνικές εποπτικές αρχές, ε, όπως γίνεται ήδη σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα συντονίσει την αξιολόγηση αυτών των ε, σχεδίων. Ο στόχος είναι οι εποπτικές αρχές να έχουν μια συνολική εικόνα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ε, ικανότητα του τραπεζικού τομέα να φτάσει τους στόχους χρηματοδότησής του. Δεύτερον, ε, η αύξηση στη συσσόρευση των ε, στοιχείων του ενεργητικού, ε, η οποία χρησιμοποιείται από τα πιστοτικά ιδρύματα για να εξασφαλιστεί η, η χρηματοπιστωτική, εξασφαλιστούν οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ε, οι επιπτώσεις είναι διτές. Από τη μία μπορεί η υπερβολική συσσόρευση τέτοιων στοιχείων του ε, ενεργητικού να δημιουργήσει μεγαλύτερες δυσκολίες για την σίγουρη χρηματοδότηση και μπορεί να δημιουργήσει πολλές προκλήσεις για την αποτελεσματική ε, διαχείριση και εποπτεία της ρευστότητας και των κινδύνων της χρηματοδότησης. Απ' την άλλη, οι πιστωτές μπορεί ε, να προσφύγουν σε άλλου τύπου στοιχεία ε, ενεργητικού σε περίπτωση που τοχεύσει το συγκεκριμένο πιστοτικό ίδρυμα. Ε, θα πρέπει να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι και γι' αυτό ακριβώς προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου συνεχή εποπτεία. Επίσης θα πρέπει τα πιστοτικά ιδρύματα να δίδουν πληροφορίες για τα, όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία Τρίτον, η ανάγκη να επεκτείνουμε τις βέλτιστες πρακτικές για να καλύψουμε τα, ε, τα καθεστώτα ομολόγων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα, τα καλυμμένα, τα, τα ομόλογα με εγγυήσεις ε, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη χρηματοδότηση των πιστοτικών ιδρυμάτων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συστήνει ε, οι αρχές αυτές να προωθήσουν την σύγκληση με βάση τα υψηλότερα τα πρότυπα. Η επόμενη σύσταση αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια για βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Έχουν ε, δημοσιεύσει συστάσεις ε, για αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια σήμερα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του σκιώδου τραπεζικού τομέα. Στην Ευρώπη ε, αντιστοιχούν σε ένα-τρει ευρώ στοιχείων που συγκεντρώνονται σε ορισμένε χώρε, κυρίω Γαλλία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. Μετά την ε, οικονομική κρίση ε, υπήρξε διεθνή συμφωνία για την ανάγκη διαθροτικών μεταρρυθμίσεων σε αυτό το τομέα. Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ε, το ESRB είναι ότι μια ενδεχομένω αποσταθεροποιητική φυγή επενδυτών για αυτά τα MMFs θα μπορούσε να οδηγήσει στη δευτερογενή επίπτωση για το ευρύτερο χρηματοοικονομικό σύστημα. Ο κίνδυνο φυγή επενδυτών μπορεί να είναι μεγαλύτερο ε, για τα αμοιβαία κεφάλαια βραχυπρόθεσμων επενδύσεων με μια σταθερή ε, καθαρή αξία, τα λεγόμενα CNAV funds, CNAV. Το Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων συστήνει ότι να είναι υποχρεωτικό για αυτά τα ε, αμοιβαία κεφάλαια να μεταμορφώνονται σε ε, ε, αμοιβαία κεφάλαια μεταβλητής καθαρής αξίας στοιχείων σε μια μεταβατική περίοδο βεβαίως. Τέλος, οι συστάσεις μας καλύπτουν και άλλες, άλλους τομείς για την μείωση του συστημικού κινδύνου που συνδέονται με αυτά τα κεφάλαια ε, ιδίω με την εισαγωγή ρητών προϋποθέσεων ρευστότητα, σε μεγαλύτερη ορατότητα και ενίσχυση της ε, υποβολής εκθέσεων και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρχών. Με τις συστάσεις της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ESRB κυρίως ε, συμβάλλει στην ανάπτυξη εύρους της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε αυτό τον τομέα. Παράλληλα, οι συστάσεις έχουν ως στόχο να στηρίξουν την παγκόσμια πρόοδο, όπως έχει πρόσφατα ε, υποστηριχθεί από το Financial Stability Board και το IOSCO από τις ε, μεγάλες οικονομίες εταίρους μας. Το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, ε, που είναι ο ομόλογος του SRB της ΕΠΑ, πρόσφατα έχει δημοσιεύσει ένα κείμενο με τον ίδιο στόχο. Τώρα, να αναφερθώ στα μελλοντικά μας σχέδια. Πρώτα απ' όλα, θα ε, στραφούμε προς τα ζητήματα διασύνδεσης ε, στο διατραπετικό σύστημα. Ένας από τους βασικούς ε, στόχους εργασίας ε, είναι να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη διασύνδεση, τα δίκτυα και τον ρόλο τους ε, σε σχέση με την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Η διασύνδεση είναι κύρια διάσταση του συστημικού κινδύνου. Όπως φάνηκε και κατόπιν της κατάρρευσης της Lehman Brothers, οι διασυνδέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων και αγορών που οδηγούν σε διαφοροποίηση σε ένα καλό περιβάλλον μπορούν να οδηγήσουν σε ε, ε, επιμόλυνση όταν υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες. Αυτό αφορά ιδιαίτερα το ESRB, καθώς η διαδικασία δημοσιονομικής ε, ολοκλήρωσης έχει δημιουργήσει πληθώρα περίπλοκων διασυνδέσεων στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού συστήματος. Μέχρι τώρα το ESRB μαζί με την ΕΣΜΑ έχει εξετάσει αυτό το θέμα σε σχέση με δύο συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, ε, συγκεκριμένα την ε, διατραπεζική διασύνδεση και την επιμόλυνση σε ό,τι αφορά την αγορά ε, των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστοτικού κινδύνου CDS. Το ESRB και η ESMA συνεργάζονται και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουν το έργο τους σε αυτόν τον τομέα δεν έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας, όμως ένα προκατακτικό ε, δίδαγμα είναι ότι μια πιο συνολική και σφαιρική διασύνδεση ε, των διασυνδέσεων μάλλον ε, του χρηματοοικονομικού συστήματος είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε πώς μεταδίδονται οι κρανασμοί στο σύστημα και πώς πρέπει να τους περιορίσουμε. Άλλο δίδυμα που θα μπορούσαμε να αντιλήσουμε είναι ότι η αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων απαιτεί έγκαιρα στοιχεία ε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς εκθέσεις ή τα λεγόμενα super spreaders. Ε, και σε τελική ανάλυση, τέτοιου είδους ανάλυση θα μπορούσε ε, να ενταχθεί στο risk dashboard του SRB και να αποτελέσει μια βάση για μια ε, σα κλίμακας επιχείρηση ελέγχου, stress testing. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι μακροπολιτικέ ε, πολιτικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ακρόαση ενώπιον τη Επιτροπή πριν από ένα χρόνο παρουσίασα τη σύσταση του SRB για την μακροπροληπτική εντολή των εθνικών αρχών. Από τότε έχει σημειωθεί ε, σημαντική πρόοδος. Αρκετές χώρες έχουν ήδη αναλάβει δράση και έχουν ε, συστήσει επιτροπές, ε, μεριτές εντολές να παρακολουθούν και να περιορίζουν συστημικούς κινδύνους. Ορισμένες από αυτέ τι χώρες, Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, κάτω χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν θέσει σε ισχύ νέα μακροπροληπτική νομοθεσία. Άλλε χώρες όπως η Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Πολωνία και Σλοβενία έχουν παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις ε, στα κοινοβούλια τους. Ε, κατανοώ ότι και άλλες χώρες έχουν αναλάβει τέτοιες ε, ενέργειες. Τέλος, άλλες χώρες που η Βουλγαρία, η Εστονία, η Ιρλανδία, Ιταλία και η Ισπανία θεωρούν ότι ήδη συνάδουν αυτή τη σύσταση. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα υποβάλουμε έκθεση στο Κοινοβούλιο στη συνέχεια. Το επόμενο βήμα στην ανάπτυξη του μακροπροληπτικού πλαισίου είναι να παράσχουμε σε αυτές τις εθνικές αρχές ένα ευέλικτο, μια ευέλικτη εργαλειοθήκη μακροπροληπτικών ε, μέσων για να διασφαλίσουμε ότι μόλις εγκαθιδρυθεί θα είναι σε θέση αυτές οι χώρες να προβλέψουν και να προλάβουν ε, την ε, αύξηση των συστημικών κινδύνων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο και σε τεχνικό επίπεδο στον αντοπισμό των ε, πρωτογενών και δευτερογενών στόχων της μακροπολιτικής πολιτικής, καθώς και ε, σε ό,τι αφορά έναν ενδεικτικό κατάλογο μέσων που ε, θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσω να αναφερθώ επιπλέον σε αυτό το ζήτημα με περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες ακροάσεις. Όπως γνωρίζετε, κάποια ε, τμήματα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, αφορούν ε, το πακέτο CRD-CRR ε, που αφορά την άμεση εμπλοκή της του ESRB στο συντονισμό των μακροπολιτικών μέτρων. Επιπλέον, ε, το προσχέδιο κανονισμού για τον SSM επίση καλεί και τον SSM να συνεργαστεί στενά με το ε, Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων. Τέλος, ε, οι δύο κανονισμοί που στηρίζουν τον ESRB θα υποβληθούν για αναθεώρηση μέχρι το τέλο του χρόνου. Σε ό,τι αφορά τι νέε θεσμικέ ε, εξελίξει, το ESRB θα βρίσκεται στην ε, διάθεση του Κοινοβουλίου ω ε, είναι απαραίτητο. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Very... ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μπορώ να σα επικαιροποιήσω για το τι συμβαίνει σε σχέση με το ESRB4. E όπου προσπάθησε το Assets Encumbrance να το θέσει το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω με επιτυχία και με την υποστήριξη του ESRB, παρόλες τις αρχικές επιφυλάξεις, νομίζω ότι θα μπορούσαν να το δεχθούν διότι θα πρέπει να μπορέσει να διασφαλιστεί ποιότητα σε σχέση με την προσπάθεια και με ιδιαίτερη σοβαρότητα για το μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Τι θα επιτρέπεται στο ESRB 4. Δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά περιοριστικό αυτό το πλαίσιο και να μην απαγορεύεται η ενδεικτική χρήση δικτών και μέσων που ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα περνάμε στο γύρο ερωτήσεων. Η πρώτη από το Ελκα, Εσείς Γκούναρ Χεκμαρκ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα δύο θέματα να αναφέρω. Αμφότερα για την ε, επίλυση προβλημάτων στο τραπεζικό τομέα και την δυνατότητα θετικής δράσης σε σχέση, σε σχέση με τις ε, ε, πλευρές κινδύνων, ένας από τους συστημικούς κινδύνους είναι ότι αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι τράπεζες σε σχέση με τη μία ή άλλη χώρα που έχουν την έδρα τους που εκτιμώντας πολλές φορές τη σημασία της σπουδαιότητα μιας τράπεζας σε μια αγορά ή τις συνακόλουθες δράσεις. Θα ήθελα να ακούσω από εσά τα σχόλιά σας, διότι προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμού στην κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Πώς βλέπετε την ισορροπία μεταξύ της χώρας υποδοχής και της αποστέλουσας χώρας. Το δεύτερο είναι κάπως ευρύτερο θέμα. Αναφερθήκατε στην προηγούμενη ακρόαση στην οποία είχατε παραστεί για τη συζήτηση για τον μηχανισμό επίλυσης ε, κρίσεων ε, και το θέμα της επίλυσης της χώρας υποδοχής και της ε, χώρας που έχει θηγατρικό υποκατάστημα σε μια τέτοια χώρα υποδοχής. Το θέμα τώρα σε σχέση με το νόμισμα θα έχουμε διαφορετικές, διαφορετικά νομίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μια ε, κατακαιρματισμένη, ε, μια κατάτμιση των δομών. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε εσείς ε, την κατάσταση και τα προβλήματα. Αντί να ε, εργαζόμαστε από κοινού σε μια κοινή βάση, να έχουμε μια τέτοιου είδους κατάτμιση. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό δεν έχω κάποιο απόφθεγμα σου ειδικό να σας δώσω για να σκεφτείτε το τι θα μπορούσατε να πείτε, αλλά θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ για την χώρα υποδοχής και τα θηγατρικά υποκαταστήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια εξάντε ε, συμφωνία για την ε, κατάσταση που θα δημιουργηθεί. Είναι ο πιο πρακτικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Για τη δεύτερη παρατήρησή σας, αυτό που προανέφερα είναι ότι οτιδήποτε και αν κάνουμε προσπαθώντας να οικοδομήσουμε αυτό το νέο μηχανισμό, η πρόθεσή μας δεν θα πρέπει να είναι και δεν θα είναι να, να υπονομεύσουμε, να καταστρέψουμε την ενιαία εσωτερική αγορά με κανένα τρόπο. Δεν βλέπω λοιπόν να υφίστανται πραγματικοί συστημικοί κίνδυνοι από το γεγονός ότι έχουμε διαφορετικές ίσως προσεγγίσεις όσον αφορά την αρχή για παράδειγμα επίλυσης κρίσεων. Ίσως όμως σε σχέση με κάποιες αναποτελεσματικότητες που θα απορρέουν, που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ενιαία εσωτερική αγορά. Αν γίνει κάτι τέτοιο αυτό θα είναι εις βάρος ε, όλων και κανείς δεν θα είναι πρόθυμος να υπομειστεί το κόστος μιας τέτοιας ε, απώλειας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και συνετοί στην κατάρτιση ε, σχεδίων για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Έχουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά Έχουμε χώρες που αυτή τη στιγμή δεν θα συμμετέχουν και δεν θα συμμετάσχουν ε, στην ε, Ευρωζώνη, στο ενιαίο νόμισμα. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σακμάκ. Το γεγονός είναι ότι η αλληλεξάρτηση μεταξύ των τραπεζών δεν ακολουθεί τα πρότυπα των ε, διαφορετικών νομισμάτων και υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος στη σουηδική περίπτωση γνωρίζουμε το τι ε, έχουμε και ποιο είναι το κεκτημένο, αλλά δεν γνωρίζουμε τι θα υπέρθει και τι θα επισυμβεί μετά. Από την, ε, τους σοσιαλδημοκράτες η Ελίζα Φερέιρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι ο μεγάλος κίνδυνος, συστημικός κίνδυνος ε, που κατέβαλε την ζώνη ευρώ είναι η εθνική υπερχρέωση, η κρατική υπερχρέωση. Αυτή τη στιγμή με την παρέμβαση που έγινε ε, με τις OMTs ε, ε, έχουμε σταθεροποιήσει την κατάσταση. Διερωτώμε όμως, αυτή θα είναι μια αρκετά ικανή λύση, αρκετά ισχυρή για να αντιμετωπιστεί το θέμα του χρέους, της χρέωσης που στο τέλος θα επιβαρύνει τα κράτη όσον αφορά τις διαδικασίες προσαρμογής. Αν όχι, τι μπορεί κανείς να σκεφτεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Δεύτερη ερώτηση, για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα ακόμα. Βρίσκεται υπό εξέλιξη η συζήτηση για την έκθεση Λικάινεν, ε, για τους συστημικούς κινδύνους. Πώς μπορεί να ε, απαμβληθούν αυτοί σε σχέση με την υλοποίηση των συστάσεων της ε, έκθεσης Λικάινεν Πώς εσείς βλέπετε να διαμορφώνονται οι ευθύνες μέσα από τον, ε, ε, την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων ε, για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Thank you. Um, the OMT... Σας ευχαριστώ. Από πλευράς OMT έχει μειωθεί ο κίνδυνος ε, ο συστημικού κινδύνου για την Ευρωπαϊκή, για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ζώνη σε σχέση με τις ε, οριστικές νομισματικές συναλλαγές. Αυτές οι νομισματικές συναλλαγές OMT ε, θα πρέπει να συνοδεύονται από σταθερές αποτελεσματικές δράσεις που θα ακολουθούν σε πολυσχηδή επίπεδα και στην νομισματική παγίωση και στον τομέα των διαθετικών ε, αλλαγών και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ε, ο συνιστός σας ε, και την δυνατότητα να μειωθεί η αναλογία της υπερχρέωσης σε σχέση με το ΑΕΠ, του βάρους του χρέους όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ. Έχουμε τις δύο πλευρές από πλευράς των δύο αυτών νομισμάτων. Η έκθεση Λίκανεν λοιπόν είναι, ο στόχος της έκθεσης Λίκανεν είναι να σχεδιάσει και να προτείνει ένα τραπεζικό πρότυπο όπου διάφοροι κίνδυνοι ιδιαίτερα επικίνδυνες ε, δραστηριότητες, ε, συστημικά τραπεζικά επικίνδυνες τέτοιες δραστηριότητες θα μπορούν να περιορίζονται. Και υπάρχει και ένα άλλο όφελος. Υπάρχει μια κοινή προσέγγιση για όλες τις χώρες που εξετάζεται μέσα από αυτή την έκθεση. Εν τω μεταξύ κάποιες χώρες ε, δραστηριοποιήθηκαν ανεξάρτητα σε αυτό το πεδίο. Η δική μου η άποψη ποια είναι. Είναι ότι σταδιακά στο τέλος τέλος θα έπρεπε να συγκλίνουμε. Να συγκλίνουμε σε μία κοινή προσέγγιση για τον περιορισμό κινδύνων από πλευρά των τραπεζών, που θα είναι κοινή προσέγγιση για όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην έχουμε διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς. Το όφελος να είναι τελικά προς όφελος όλων, να μην αποβεί βάρος ε, της ε, ενιαίας ε, εσωτερικής αγοράς μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αυτή η προσέγγιση. Η δική μου όμως άποψη είναι ότι ευελπιστώ ότι θα συγκλίνουμε τελικά σε κοινού κανόνες και κανονισμούς για να περιορίσουμε αυτούς τους κινδύνους σε τέτοιου είδους δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς θα θέλατε να επανέλθετε παρακαλώ κυρία Φερέιρα. Όταν κάνετε λόγο, όταν κάνετε λόγο για την ανάπτυξη, η ανάπτυξη φαίνεται ότι είναι κυρίαρχη, ας το πω έτσι, κυρίαρχη συνιστόσα σε όλα όσα κάνουμε και συζητούμε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να στρέψουμε την, την προσοχή μας στις αγορές όπου, υπάρχει η προοπτική τέτοιας ανάπτυξης και σε σχέση και με τις ισοτιμίες, οι συναλλαγές. Έχετε κάποια δυνατότητα να μας πείτε σε σχέση με την ισοτιμία του ευρώ τι μπορεί και πρέπει να γίνει ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν τις εξωτερικές αγορές για τη δική τους εσωτερική ανάπτυξη από τη ζώνη ευρώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντράγκη, σας ευχαριστώ. Επισημαίνει το ότι πιέζει ο χρόνος η πρόεδρος Σύντομα, η ισοτιμία, η νομισματική ισοτιμία είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την νομισματική σταθερότητα. Θα έχουμε νέες προβλέψεις και προοπτικές ε, πολύ σύντομα για την ισοτιμία του ευρώ. Ξέρουμε και εδώ δεν ομιλώ από πλευρά ε, του, του SRB αλλά ως, υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρέπει να δούμε τώρα στο εύρος μακροπρόθεσμα των ισοτιμιών του ευρώ το θέμα της ε, νομισματικής σταθερότητας και πρέπει αυτό να ληφθεί κυρίαρχα υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σιλβί Γκουλάρ για την Άλντε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Στη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής του ESRB για το SSM, για το ε, νέο εποπτικό μηχανισμό, στην παράγραφο 6, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες. Έχετε την αίσθηση ότι το άρθρο 5 του σχεδίου του SSM είναι παρκές, σας επιτρέπει δηλαδή να εντοπίσετε τις περιπτώσεις και να ενημερώσετε την ΕΚΤ για, τις, για τις περιπτώσεις που χρήζουν ε, εποπτείας. Μερικές φορές εσείς εποπτεύετε, μερικές φορές οι εθνικές ε, εποπτικές αρχές. Ε, αν έχετε ειδικά, ειδικές παρατηρήσεις να κάνετε, εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια και θα ήθελα να τις ακούσω για, το, για την έκθεση αυτή που θα ετοιμάσουμε για, το, για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Δεν έχω να σας, ειδικά σχόλια να σας κάνω για το κείμενο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Είναι ένα σημαντικό βήμα που θέλω να... Αυτό θέλω να πω. Αυτό το βήμα το έχουμε πάρει όλοι μαζί, το έχουμε κάνει όλοι μαζί για να προχωρήσουμε προς μια πιο γνήσια και πραγματική νομισματική ένωση. Ε, το βήμα αυτό θα είναι σημαντικό αν είναι μεγάλο. Θα πρέπει να έχουμε ισχυρή εποπτεία. Δεν θα πρέπει να είναι ένας τρόπος για να, καλύψαμε, να καλύψουμε τις αδυναμίες ε, και οι αδυναμίες αυτές θα παραμείνουν. Όχι, θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στην εθνική εποπτεία και στην ευρωπαϊκή εποπτεία, την κεντρική. Αλλά η κατάσταση πρέπει να αλλάξει ούτως ή άλλως. Και αυτό το είπα από την αρχή. Έχω την αίσθηση ότι το SSM δεν είναι σαν ένα είδους κέικ όπου το μοιράζουμε και λέμε «Α, αυτό το κομμάτι ας πούμε γίνεται στη Φραγκφούρτε και το υπόλοιπο σε εθνικό, ε... σε εθνικό επίπεδο». Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι τμήμα του μηχανισμού, τμήμα του ΚΕΙ και όλοι μαζί κάνουμε αυτή την εποπτεία. Και στο κέντρο και σε εθνικό επίπεδο κάνουμε εποπτεία. Επομένως, η αρχιτεκτονική θα πρέπει να εμπλέξει όλους τους εταίρους και όλοι οι εταίροι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί. Οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν όχι μόνο τη γνώση, αλλά και την παράδοση και την, τις εξουσίες για να είναι αποτελεσματική σε εθνικό επίπεδο. Αν όμως, αν ε, η δουλειά που κάνουν οι εθνικές εποπτικές αρχές ε, δεν γίνεται και δεν καλύπτεται ας πούμε και από την, το την κεντρική εποπτεία που ασκείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε θα έχουμε χάσει τη, το τρένο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να θέσω μια ερώτηση. Έχω μια πολύ εξειδικευμένη ερώτηση για την αναδιάρθρωση και την ανακεφαλαιοποίηση των μη φερέγγιων τραπεζών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι μια πρακτικού χαρακτήρα ερώτηση, αλλά έχει επιπτώσεις και σε άλλα θέματα εξίσου επίσης. Δημιουργώντα είτε ένα καλό είτε ένα κακό προηγούμενο βάσει αυτό. Στην περίπτωση τη Ελλάδα οι τέσσερι μεγαλύτερε τράπεζες όχι μόνο έχουν πολύ αρνητικά από πλευράς τραπεζικού ε, στοιχείου ε, περιουσιακά στοιχεία, αλλά έχουν και θετικά στοιχεία και πρέπει να επιληθεί αυτό το πρόβλημα και να ε, εξηγιαθεί το ε, περιουσιολόγιο τους ε, και να υπάρχει λιγότερη ανακεφαλαιοποίηση εις βάρος των φορολογουμένων που θα πρέπει να λειτουργήσει. Έχουν μια ολόκληρη αυτοκρατορία στα Βαλκάνια ελληνικές τράπεζες, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στη Μακεδονία, Αλβανία και είναι αυτές που έχουν, αποκομίσουν τα μεγαλύτερα κέρδη έχουν καλύτερες επιδόσεις από τις άλλες τράπεζες. Γιατί δεν θα μπορούσαν λοιπόν να πωλήσουν αυτά τα ε, περιουσιακά του στοιχεία και να χρειάζονται πολύ λιγότερα χρήματα από τους φορολογούμενους στο εσωτερικό της Ελλάδας για την εξυγίανσή τους. Οι κυπριακές τράπεζες είναι σε χειρότερη κατάσταση. Όχι μόνο δεν υπάρχει φερεγγιότητα, δεν υπάρχει ρευστότητα, αλλά είναι πολύ πιεστικά τα προβλήματα. Είναι παραπλανητικά ωστόσο αυτά τα οποία τίθενται συζήτηση. Είτε θα υπάρξει πλήρης ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είτε όχι. Τότε γιατί δεν ξεκινάμε μία αντιμετώπιση όλων των τοξικών αυτών στοιχείων και να κλείσουν οι τράπεζες αν θα έπρεπε στο τέλος. Το αγγλο-ιρλανδικό παράδειγμα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Προσπαθήσω, δεν ξέρω πόσο μπορώ να είμαι πλήρης ε, για το θέμα της Κύπρου, γιατί έχουν, ε, δεν έχουν τελειώσει οι συζητήσεις και δεν θέλω να προδικάσω τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν ε, χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τις ελληνικές τράπεζες. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η, η Τράπεζα της Ελλάδος ετοίμασε την έκθεση για την ανακεφαλαιοποίηση με όλα τα νούμερα για όλες τις τράπεζες και τις ε, εξατομικευμένες ανάγκες. Θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το τέλος Απριλίου του 2013 οι τράπεζες αυτές. Έτσι του ζητείτε από την Τράπεζα Ελλάδος. Αν είχαν αυτά τα περιουσιακά, τα περιουσιακά στοιχεία, αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού εμπασχεπτώσει, σίγουρα θα ληφθούν υπόψη, ούτω ώστε να υπολογίσουμε το λόγο κεφαλαίου τους. Για τις βασικές τράπεζες, ε, που είναι στη δεύτερη φάση ανακεφαλαιοποίησης ε, για να, έχουν, ε, να φτάσουν σε ένα επίπεδο 9% του CT1 και μετά την επιπρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση για τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες η φερεγγιότητά τους έχει αποκατασταθεί. 57 εκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια ευρώ πήγανε για πολιτικές ε, νομισματικού χαρακτήρα. Έχει γίνει πρόοδος, δηλαδή το, το ποσοστό του, της, βοήθειας, ε, κατε, της κατεπήγουσας βοήθειας που πρέπει να δώσουμε και με αυτή την επιχείρηση που κάναμε στην Ελλάδα και την Ιρλανδική συμφωνία μεταξύ της, Ευρωπαϊκής, της Ιρλανδικής Κεντρικής Τράπεζας και της ε, κυβέρνησης, το ποσό του, που δίνουμε για τον κατεπήγοντα δανεισμό έχει μειωθεί σημαντικά. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Πάμε τώρα στην ΚΟΕ. Τον κύριο Χουντή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση συμπτωματικά μοιάζει να αφορά την Ελλάδα. Αλλά θα δείτε ότι έχει μια γενικότερη σημασία και όπως και οι συνάδελφοι. Παρακολουθείτε, διότι νομίζω ότι είσαστε υποχρεωμένος, τη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά από δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρτ και κορυφαίων οικονομολόγων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ήταν λάθος, διότι έγιναν λάθος υπολογισμοί και ε, μπαρδεύσαμε τους πολλαπλασιαστές. Προχτές ο κύριος Ρεν κοινοποίησε στους Υπουργούς Οικονομικών των χωρών των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εσά, έτσι λέγεται, επιστολή που λέει ότι αυτή η υπόθεση με τους πολλαπλασιαστές έχει περιορισμένη δράση και επομένως πρέπει να σταματήσει η συζήτηση. Φυσικά τα αποτελέσματα μιας τέτοιας λάθος επιλογής υπολογιστών δεν θα τα παριθμίσω, τα γνωρίζουμε. Η ερώτηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι το μόνο πια μέλος της Τρόικα που δεν έχει μιλήσει με σαφήνεια σχετικά με το θέμα των πολλαπλασιαστών. Σας ρωτώ, και έχει τη γενικευμένη σημασία, διαθέτετε την τεχνογνωσία ή την έχετε εκχωρήσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μου απαντήσετε αν αυτές οι μελέτες για τους πολλαπλασιαστές στην περίπτωση της Ελλάδας ή και γενικότερα είναι σωστές ή λάθος προλογικά την παρατήρηση είναι περισσότερο για τον πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το ερώτημα και όχι για το ESRB. Θα απαντήσω όμως, συμφωνώ απόλυτα με τον Όλι Ρεν και την Κριστίν Λαγκάνσα όσα είπαν. Πολλές συζητήσεις έγιναν για κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να είχε αξιολογηθεί με απόλυτη βεβαιότητα εκ προημίου. Και θα ήθελα να σας αναγνώσω το εξής παράθεμα. Όσον αφορά του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστές πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι οι κυριότεροι λόγοι για την μεγαλύτερη ύφεση δεν, βρίσκονται στους πολλαπλασιαστές αλλά στο, στη φύση αυτού του προγράμματος και σε κάποιες καθυστερήσεις υλοποίηση του προγράμματος ε, που περιόρισαν την αποτελεσματικότητα και σε σχέση με το 15% του ΑΕΠ το 2009 υπήρξε απώλεια της αγοράς και υπήρξε ναι, μεγάλη ανάγκη δημοσιονομικών προσαρμογών. Σαν συνέπεια όλων αυτών μειώθηκε το πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής και παρατάθηκε το χρονικό πλαίσιο κατά δύο έτη. Οι πιστωτές διευκόλυναν την Ελλάδα παρέχοντας αυτή τη διευκόλυνση. Πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι το αναθεωρημένο πρόγραμμα ανταποκρίνεται με την επικαιροποίηση της οποίας έτυχε ήδη τον Ιανουάριο. Νομίζω ότι αυτό απαντά πλήρως στο ερώτημά σας. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο να τα αναθεωρήσουμε όλα αυτά, ακόμα και το πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Το κλειδί για την επίλυση της κρίσης εξακολουθεί να είναι στα χέρια της Ελλάδας. Και προσβλέπουμε στο ότι η κυβέρνηση θα πρέπει πλήρως να, προσα... να συμμορφωθεί με το πρόγραμμα στην υλοποίησή του. Αυτό νομίζω εξαντλεί το θέμα των πολλαπλασιαστών, των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών. Υπήρξε μια έντονη και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και μεταξύ των οικονομολόγων και των στελεχών και στην, ε, στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να εξεταστεί πλήρως και εξαντλητικά το θέμα των πολλαπλασιαστών και να υπάρξει μια τελική συμφωνία. Γι' αυτό το θέμα τώρα, σε αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει η αξιολόγηση των πραγμάτων την οποία κάναμε για την κατάσταση τη Ελλάδα. Ευχαριστώ. Και τώρα σε σχέση με το έργο σας από πλευρά σε ESRB, σε αυτή την ακρόαση, σε αυτό θα πρέπει να εστιαστούμε και να δούμε την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων από πλευρά αυτής της προοπτικής. Ευχαριστώ. Ε, Μοργάντη, ευχαριστώ. Είμαι από την Τοσκάνη. Ε, η τράπεζα Μόντε Διπάσκη, που είναι η πιο παλιά τράπεζα και που βρίσκεται σε δυσχέρεια. Τα περισσότερα προβλήματα της τράπεζας αυτής οφείλονται σε αγορές που έγιναν ε, το 2007. Ε, πολύθηκε η Άντων Βεν και η Σανταντέρ. Το βασικό πρόβλημα των συναλλαγών αυτών οφειλόταν στο ότι η τη Πάσκη δεν είχε λεφτά για αυτή την αγορά που έκανε, την εξαγορά που έκανε. Και όποιος έλεγε αυτή την συναλλαγή θα έπρεπε να έχει εμποδίσει αυτή τη συναλλαγή. Πώς εκτιμάτε αυτή την εκτίμηση εσείς. Και γιατί ο τότε διοικητή της Τράπεζας Ιταλίας δεν μπλόκαρε αυτή την συναλλαγή. Είναι σωστή αυτή η υπόθεση ότι δεν έπρεπε να γίνει συναλλαγή. Επίσης, ε, η μία από τις δύο τράπεζες που εξαγοράστηκαν από τη Μόντε Πάσκη ε, εξαγοράστηκαν σε πολύ ψηλότερη τιμή από ό,τι έπρεπε. Η Goldman Sachs ασχολήθηκε με την συναλλαγή μεταξύ ε, Τράντον Βένετε και μία Ολλανδική τράπεζα το 2005 όταν έπαιζε... Εσείς τότε είχατε σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό της Goldman Sachs. Ε, η τιμή που πληρώσαμε στο Santander το 2007 δεν ήταν υπερβολικά ψηλή και ίσως ε, έκρυβε και κάποιες λαθροχειρίες. Δεν συμφωνείτε με αυτό? Σας παραπέμπω στη δήλωση που έκανε η Banca d'Italia στην ιστοσελίδα της. Η Banca d'Italia έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να εξασφαλίσει ότι υπάρχει λογοδοσία και υπάρχει και ένας λογαριασμός, μια λογοδοσία στην ιστοσελίδα της Banca d'Italia. Η προκαταρτική γνώμη του Δούνου του είναι ότι η Τράπεζα Ιταλίας ε, πήρε έγκαιρη και κατάλληλη δράση. Αυτό είπε του Δούνου του, εντός των πλαισίων του νομικού ρόλου της για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Υπήρξε εποπτεία στενή εποπτεία και η αντίδραση, η εποπτική αντίδραση ε, κλιμακώθηκε ε, όπως έπρεπε καθώς το πρόβλημα οξύνθηκε. Και συνεχίζει στο ίδιο, στον ίδιο τόνο. Σας παραπέμπω λοιπόν σε αυτά τα δύο έγγραφα. Το ένα της Banca d'Italia που υπάρχει στην ιστοσελίδα της και το άλλο, ε, το δεύτερο ήταν δήλωση του Δουνουτού. Και μην ξεχνάτε ότι εγώ έστειλα αυτές τις δύο αποστολές εποπτείας ε, στις τράπεζες αυτές. Εγώ ήμουν υπεύθυνο. Ευχαριστώ. όπω είπα πριν, θα πρέπει να επανέλθουμε στα ζητήματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων. Ξέρω ότι υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα, όμως εδώ θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα που αφορούν το ESRB. Νομίζω όμω ότι ξέφυγαν από αυτό το θέμα τα δικά σα ερωτήματα, συνάδελφε. Νομίζω ότι απαντήθηκαν μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση. Μια επερώτηση. Για την ESRB ναι, αλλά πολύ γρήγορα. Μόνο. Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω για το Monte Τιπάσκι. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Όχι. Για... Όχι, την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Και δεν είναι θέμα του ESRB εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ESRB. Όχι, συγγνώμη. Ο Βέρνερ Λάγκεν θα πάρει το λόγο. Απόλυτα για αυτό το θέμα τώρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την περιγραφή των μέτρων από πέρυσι. Κατά το παρελθόν επανειλημμένα μιλήσαμε και μιλούσαμε για την κρατική υπερχρέωση. 13 δις ευρώ, σχετικά υψηλή. Όμως η ακαθάριστη υπερχρέωση ε, των παθητικών μείων του ιδίου κεφαλαίου είναι υψηλότερο ακόμα ποσό, 31 δις ευρώ από αυτά 9,2 δις στις χώρες κρίσης. Το θέμα είναι πώς θα διεφύγουμε, θα διεξέλθουμε από αυτή την κρίση. Αναφέρατε αρκετά παραδείγματα. Το πιο σημαντικό είναι η αύξηση των ποσοστών ιδίων κεφαλαίων και βρισκόμαστε σε διαβούλευση και υποδιαπραγμάτευση. Σύμφωνα με μια μελέτη του ΩΣΑ, 110 δις ευρώ θα χρειαζόντουσαν επιπρόσθετα για αυτά τα κεφάλαια. Σε ποιο χρονικό διάστημα θεωρείτε εσείς αυτό ως πρόεδρος ε, του ESBR εφικτό και ποια μέτρα θα, ήταν, ε, θα είχαν νόημα να αναλυθούν. Αναφέρατε τις σκιώδεις τράπεζες. Τρεις χώρες αναφέρατε. Γαλλία, ε, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο. Και είπατε ότι, και αναφέρατε και τα, τα θέματα του Ταμείου και της, ε, των, των ε, δράσεων. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις σχετικά. Και τρίτος τομέας, πώς βλέπετε τον ε, διεθνή συντονισμό στα θέματα περιορισμού κινδύνων, συστημικού, συστημικών κινδύνων. Ευχαριστώ. Για την πρώτη σας ερώτηση η έναρξη σε ισχύ του, της Βασιλείας 3 της Συμφωνίας προχωρεί. Και σωστά γίνεται αυτό, διότι οι ρυθμιστές ήθελαν να αποφύγουν αρνητικές επιπτώσεις ε, στη μακροοικονομική κατάσταση που ήδη ήταν αποδυναμωμένη η κατάσταση πραγμάτων μακροοικονομικά. Θα αξιολογηθούν αυτά κατά την εξέλιξη αυτού του έτους. Θα αξιολογηθεί η ποιότητα των ε, στοιχείων αυτών και των διαφορετικών τραπεζών η ποιότητά τους. Μέχρι σήμερα οι τράπεζες ε, συνέλεξαν κεφάλαια και μέσα στην ε, κεφαλαιοποίηση όσον αφορά αυτό το καθεστώς ε, έγιναν τέτοιες δράσεις για την διασφάλιση, συλλογή κεφαλαίων και όχι τόσο την απομόχλευση. Θα αξιολογήσουμε την κατάσταση μέχρι τα τέλη του έτους. Η επόμενη ερώτησή σας ήταν για τα ταμεία και την διάθεση κονδυλίων από αυτά τα ταμεία. Γι' αυτό το, για αυτή τη συνιστόσα μάλιστα έχουμε διάφορες δράσεις και στοιχεία τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη. Ο συντονισμός αναφέρεται στον κύριο Ντράγκη. Συντονισμός. Μάλιστα. Όσον αφορά τον συντονισμό τώρα με τις αρχές ε, των ΙΠΑ ενημερωνόμεθα και επικαιροποιούμεθα για τις συζητήσεις ε, που ε, διεξάγονται. Υπάρχουν επαφές ε, στο επίπεδο στελεχών και αξιωματούχων και υπάρχει και μια διακριβωτική αποστολή από πλευράς αριθμιστών για παράδειγμα. Μπάφιν για παράδειγμα που προείδρευσε αυτών των εργασιών και που κατά την, τις αρχές Μαρτίου θα υποβληθούν συστάσεις και συμπεράσματα από πλευράς τους. Σε παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Υπάρχει έγγραφο της ε, Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας, Fed, Κεντρικής Τράπεζας ε, των ΗΠΑ, σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι αν μπορώ να το πω, είναι πιο προηγμένο στις δικές μας συστάσεις. Έχουμε προχωρήσει πιο πολύ από αυτά τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση στη ΣΥΠΑ σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στη ΣΥΠΑ και να προχωρήσουν και εκείνοι περαιτέρω. Μια σύντομη επερώτηση Ήδη έχουμε συζητήσει για την μηδενική αξιολόγηση, το μηδενικό επίπεδο των κρατικών ομολόγων. Τώρα ένα δις είναι εκείνο το οποίο διατίθεται και ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη το ποσοστό αυτό, η διαφορά επιτοκίου χρησιμοποιείται ώστε περισσότερα ακόμα να επιτευχθούν. Στόχος είναι μέσω της τραπεζικής εποπτείας η κρατική χρηματοδότηση να διαχωριστεί σε σχέση με την τραπεζική ε, κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν συμμορφώνονται στο Νότο. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω για τη μηδενική αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα από τα θέματα το οποίο θα αναμέναμε να συζητηθεί στην, στο Γενικό ε, Διευθυντικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι μακροπρόθεσμες προοπτικές λύσεων όλα αυτά και απαιτήσει αυστηρότερες για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα για την επίλυση της κρατικής υπερχρέωσης. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ένα τέτοιο μηδενικό επίπεδο με την ε, ενιαία, ας το πω διάσταση ή να υπάρξει και μια διαφοροποίηση. Ή θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και πολυμορφοποίηση των απαιτήσεων αντίστοιχη προσαρμογή των τρίτο πυλώνα όσον αφορά τις απαιτήσει για αποκάλυψη στοιχείων και δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων και διασφάλιση ώστε να μπορέσει η έκθεση κινδύνου να μπορέσει και εκείνη να καλυφθεί σε σχέση με τις διατάξεις που θα ισχύουν. Μπορείτε να δείτε ότι εξετάζουμε λοιπόν πολυσχηδώς διαφορετικά μέτρα και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα πολύ περίπλοκο πλαίσιο αυτό, ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Πρέπει να εισαχθούν όλα αυτά με μια συγκεκριμένη χρονική προοπτική όσον αφορά τη χρονική συνιστόσα. Έχουμε όμως διάφορες ε, εναλλακτικές δυνατότητες. Ε, το ESRB γνωρίζει απόλυτα τις συστημικές επιπτώσεις που συνέχονται από αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Πολλά θα πρέπει να γίνουν λοιπόν σε σχέση με τα κράτη-μέλη και τις συζητήσεις όταν θα έρθει η ώρα να υποβάλει και το Κοινοβούλιο προτάσεις ή τροπολογίες από πλευρά τους και σε σχέση και με τις ε, ε, ε, διάφορες εξαιρέσεις όσον αφορά το άρθρο 145 για παράδειγμα του CRR διότι σίγουρα ο κίνδυνος του κρατικού χρέους πρέπει και αυτός να αντιμετωπιστεί και ίσως θα μπορούσε, ας το πω έτσι, να υπάρξει μια εξειδικευμένη προσέγγιση για αυτή την προοπτική. Ίσως θα μπορούσε έτσι να υπάρξει μια προσαρμογή, διόρθωση, ώστε να μπορέσουμε μέσα στο πλαίσιο της, Βασιλείας, ε, της Συμφωνίας της Βασιλείας να προχωρήσουμε. Εσείς κύριε Ντόφαν, στη συνέχεια έχετε τον λόγο. Θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να ε, θέσω την εξής ερώτηση σε εσάς, λέει ο κύριος Ντόφμαν. Εδώ στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή σε σχέση και με τους συμψηφισμούς ή της, ε, την επίλυση των προβλημάτων. Κυρίως αντιμετωπίζουμε το θέμα των CSDs και θα πρέπει να λάβουμε αυτή την πτυχή υπόψη σε σχέση με τις τραπεζικές δραστηριότητες και την λειτουργία αυτών των μέσων. Είναι επικοδομητικό να υπάρξει διάθεση ε, ρευστότητας, να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Θα μπορούσε να ε, διασφαλιστεί αυτό μέσα στο πλαίσιο αυτό ή πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Η πλειοψηφία των μελών της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής ήταν υπέρ του να συνεχίσουμε την προσπάθεια συμβίωσης ε, μέσα στο CST με τις ε, τραπεζικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση να υπάρχει έγκριση στο ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτές τις δράσεις. Ερώτηση που θα ήθελα να σας απευθύνω. Πώς βλέπετε εσείς τον ρόλο λοιπόν του ESRB μέσα σε αυτές τις προοπτικές. Στο ρυθμιστικό ρόλο αυτών και ιδιαίτερα τι θα μπορούσε να γίνει για παράδειγμα για να υπάρχουν οι αναγκαίες εγκρίσεις στον τραπεζικό τομέα λυπούμε το ESRB δεν ε, ε, έχει ασχοληθεί ακόμα με αυτό. Είναι κάτι το οποίο ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, επομίζεται αυτή, αυτού του θέματος. Γραπτός θα μπορούσα να σας διαθέσω μια απάντηση, να σας διαβιβάσω την απάντησή μας, αλλά θα είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ασχολείται το ESRB με αυτό. Μάλιστα, επανερχόμαστε λοιπόν στο θέμα μας. Θέλετε να επανέλθετε εσείς ε, κύριε Ευρωβουλευτά, όχι. Τώρα λοιπόν οι σοσιαλδημοκράτες, Ούντο Μπούλμαν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα αν γίνεται να επανέλθω στο πακέτο ε, στις δεσμες μετρων μέτρων C4 και ε, μας έχει απασχολήσει και η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτή αυτό το πακέτο μέτρων αρχικά υπέβαλε την πρόταση άσχετα το τι θα γίνει με την αξιολόγηση των ε, κρατικών ομολόγων στο μέλλον τα ευρωομόλογα να έχουν ε, την μηδενική αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο θεωρούμε θετικό αλλά και σε σχέση με το, την ομάδα του ΕΛΚ και το συνάδελφο Βέρνερ Λάγκεν να πω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στραφούμε δύο θέματα βρισκόμαστε στην τελική φάση αυτού του πακέτου μέτρων Εξακολουθεί η συζήτηση για τα μέσα ρευστότητας και υπό το πρίσμα νέων συζητήσεων σε σχέση με τα θέματα βασιλείας κάλυψη ε, των θεμάτων ρευστότητας που θα πρέπει να επεκτείνεται σε αυξημένες απαιτήσει ώστε ε, να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είναι όλα αυτά σωστά. Θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε όσον αφορά τις ε, ρυθμίσεις ε, της Συμφωνίας Βασιλείας ή μήπως θα έπρεπε να απόσχουμε από τέτοιες ε, ας το πω χαλάρωσης και να είμαστε πιο αυστηροί, να αυστηροποιήσουμε περισσότερο τον τομέα αυτό. Από την άλλη πλευρά έχουμε και το θέμα της ελαστικοποίησης, να υπάρχει δυνατότητα για κάποιες χώρες να εκμεταλλευτούν μια τέτοια δυνατότητα, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους όσον αφορά τις κεφαλαιακές αγορές, ε, τις κεφαλαιακές τους ανάγκες. Άλλοι Άλλες χώρες επιμένουν στο να υπάρξουν κοινοί κανόνες και κανονισμοί όσον αφορά μια κοινή οργάνωση αγοράς και δεν θέλουν να υπάρξουν πόρτες και παράθυρα για εξαιρέσεις. Εσείς υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου της, του ESRB πώς βλέπετε μια τέτοια προοπτική και ποια θα ήταν η μορφή μιας τέτοιας ρύθμισης. Μικρόφωνο. Την πρώτη σας ερώτηση για το CRD. Νομίζω ότι η τελευταία συμφωνία της Βασιλείας για το θέμα αυτό είναι μια καλή συμφωνία ουσιαστικά. Θα μπορούσα να πω ότι όλα όσα έπρεπε να αναφερθούν αναφέρθηκαν τότε και διατυπώθηκαν από τον, προ, τους προέδρους των Αρχιών κρατών και ε, κυβερνήσεων και δεν έχω κανένα λόγο να διαφοροποιηθώ όσον αφορά αυτές τις τοποθετήσεις. Ουσιαστικά η συμφωνία αυτή αξιολόγησε και στάθμισε την πραγματικότητα του χώρου της Ευρωζώνης και της κατάστασης των τραπεζών σε αυτήν και πώς οι ρυθμίσεις για την ρευστότητα θα είχαν επιπτώσεις στα πρότυπα για τη λειτουργία αυτών των τραπεζών. Να μην ξεχνάμε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η διατραπεζική αγορά δεν μπόρεσε να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι τράπεζες αύξησαν την εξάρτησή τους από την κεντρική τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το γεγονός είναι ότι η δανειοδότηση, η άντληση κεφαλαίων και η διάθεση των κεφαλαίων αυτών σε δάνεια και πιστώσεις δημιουργούσε απώλειες σε αυτές τις τράπεζες. Η Συμφωνία της Βασιλείας λαμβάνει υπόψη αυτή την κατάσταση και προσπαθεί να τροποποιήσει τα θέματα ρευστότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει η συμφωνία αυτή να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς να επιβάλλει κυρώσεις ε, ε, στα τραπεζικά ιδρύματα σε σχέση με τη λειτουργία τους όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ευρύτερη συνένεση από πλευρά ESRB ότι δεν θα πρέπει να ανεχόμαστε μια πολιτική χαλάρωσης όπου ένας ε, μια χώρα θα την καλύτερη καλύτερη αντιμετώπισης από μια άλλη. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν σε ένα συντονισμό των πολιτικών μας να διασφαλίσουμε αυτές τις αρχές. Η e SRB από κοινού στο έργο αυτό για τον συντονισμό από με την CRD-CRR θα μπορεί να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο στις δράσεις και αποφάσεις τους. Να εξεταστεί το πλαίσιο αυτής της τραπεζικής πολιτικής με ε, γνώμονα και την ε, ε, ενιαία εσωτερική αγορά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έχουμε έναν ευέλικτο και γόνιμο διάλογο με τις εθνικές αρχές, με τη, πάντα με βάση τις ανάγκες συντονισμού, ώστε να αποφύγουμε αρνητικά φαινόμενα. Συντονισμό λοιπόν προβλέπεται και έτσι η ESRB θα διαδραματίσει ένα συντονιστικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστούμε πολύ και με αυτό ολοκληρώνουμε την ακρόαση για το ESRB Ακριβώ στα χρονικά μας όρια. Ο επόμενος νομισματικός μας διάλογος θα είναι στι 8 Ιουλίου για συναφή θέματα. Παραμείνετε στις θέσεις σας, στα έδρανά σας για ένα λεπτό, διότι ο Αντιπρόεδρος Παύλο θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις ε, και θα, θα συνοδεύσει τον ε, κύριο ε, Ντράγκη εκτός αίθουσας, θα επανέλθει. Να μείνετε στις θέσεις σας παρακαλώ. Hello, everyone. We'll take a few... Ένα μικρό διάλειμμα, αλλά τέλος πάντων, για να περάσω στις ανακοινώσεις ε, του Προέδρου στις 19 ε, Φεβρουαρίου, αύριο δηλαδή, θα υπάρξει μια αλλαγή της αίθουσα συνεδρίασης. Στην αίθουσα ASP 5G3 θα συνεδριάσουμε. λόγω της σημερινή ε, συνεδρίασης και της συνάντησης με τον κύριο Ντράγκη θεωρήθηκε πιο κατάλληλο να συνεδριάσουμε εδώ σήμερα. Για τους ε, τριμερείς ε, διαλόγους στις 5 και 6 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο έλαβαν χώρα τέτοιοι διάλογοι και θα συνεχιστούν μέσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα για προετοιμασία για τα ζητήματα όπως ε, Βασιλεία 1. Ορισμός ε, επενδυτικών επιχειρήσεων και διευθετήσεων για την ε, αξία για την έκθεση των κεντρικών συμβολωμένων. Για την τραπεζική εποπτεία ε, υπάρχουν ε, προτάσεις ε, τροπολογιών για όλα τα πολιτικά θέματα και είναι επιτάπητος όλα τα μέρη που εμπλέκονται θα πρέπει να αποτιμήσουν ότι έχουμε επιτύχει. Ο επόμενος πολιτικός διάλογος, τρίλογος μάλλον, θα λάβει χώρα αύριο. Για το φισκάλης ο πρώτος διάλογος για το πρόγραμμα Φισκάλης έγινε στις 13 Ιανουαρίου. Κάποια πρόοδος έχει γίνει στους εξής τομείς. Συμμετοχή ε, των φορολογουμένων τρίτων χωρών σε κοινέ δράσεις και δράσεις ε, κατάρτισης και ανθεκτικότητα του προϋπολογισμού. Έχουν γίνει τεχνικές δουλειές σε διάφορα επίπεδα. Ε, στις 20 ε, Φεβρουαρίου θα γίνει μια τεχνική συνάντηση. Ο επόμενος τρίλογος θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου με σκοπό να δει τις προτεραιότητες και να κάνει μια παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, ο, έκτης, ο έκτος τρίλογος ε, έγινε στις 6 ε, Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Ε, έχει σημειωθεί περαιτέρω πρόοδο σε διάφορα άρθρα στο θέμα του ECB. Τα περισσότερα πολιτικά θέματα έχουν εντοπιστεί ε, η πρόοδος έχει γίνει και στα πιο τεχνικά θέματα. Ο επόμενος τρίλογος θα γίνει στην, ε, στις 21 Φεβρουαρίου και θα αντιμετωπίσει την το θέμα της, ε, του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Οι διαπραγματεύσεις για την αρχή είναι για την αρχή αυτή, την τραπεζική αρχή, είναι σε αρχική φάση. Και το τελευταίο σημείο είναι η υιοθέτηση το αναθεωρημένο χρονοδιαγράμματο του 2013 για τις συνεδριάσεις τη Επιτροπής. Μετά την υιοθέτηση που έγινε ε, στην Ολομέλεια για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών και μετά από την πρόταση που έγινε, έγινε από, την, από τους Προέδρους θα βρείτε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων του 2013. Η αλλαγή είναι ε, στις 9 και 10 Οκτωβρίου, τέσσερις μισές μέρες, η εβδομάδα 21 Προβλέπετε τώρα να, ε, εκεί να λάβει χώρα η Ολομέλεια του Οκτωβρίου. 24 Σεπτεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και 3 με 6.30 το απόγευμα. Και τη Δευτέρα 13 ε, Σεπτεμβρίου, μόνο το απόγευμα, 3 με 6.30. Δευτέρα 13 Οκτωβρίου από τις 3 με 6.30. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θα θεωρήσουμε ότι αυτό το σχέδιο χρονοδιαγράμματος έχει υιοθετηθεί. Δεν έχετε σχόλια, άρα αυτό υιοθετήθηκε. Τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο στις 9 η ώρα το πρωί θα τα ξαναπούμε στην αίθουσα 5G3.